colleagues i would like to open the meeting of the subcommittee on human rights and we hope that there will be a flow of members to this meeting very soon because we have an Πάρα πολύ ενδιαφέρον το απόγευμα που μπροστά μας γιατί έχουμε δύο, δύο θέματα να συζητήσουμε πρώτα πρώτα την τεχνολογία των νέων μέσων ενημέρωση των νέων τεχνολογιών δυνατότητε, κίνδυνοι, καινούριο θέμα, ενδιαφέρον. Έχουμε πάρα πολύ εξαιρετικού προσκεκλημένου να μα μιλήσουν και γι' αυτό είπαμε στη συνέχεια συζητήσουμε το Freedom House για το πώς έχει κατάσταση για τι μεταρρυθμίσει και τα ανθρώπινα δικαιώματα στον αραβικό κόσμο. Στις 5.30 θα αρχίσει αυτό το τελευταίο θέμα. Για να δούμε, γίνανε πολλά από τότε που τα είπαμε για τελευταία φορά και γι' αυτό και θα σας κάνω την εξή ανακοίνωση. Να σας ε, αναφέρω ότι στις 10 Ιουνίου θα έχουμε εκτακτή συνεδρίαση. 9 η ώρα. Θα συναντηθούμε με τον Ισπανό πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για να συζητήσουμε διεξοδικά τα θέματα σχετικά. Τι έγινε από την αρχή του έτους. Και όπως είπαμε προηγουμένως, θα κάνουμε την ίδια μέρα αυτό που αναλύθηκε σήμερα, δηλαδή τη συνεδρίαση του διευρυμένου Προεδρείου, γιατί ε, πάρα πολλοί συνάδελφοι που θα έπρεπε να συμμετάσχουν ήταν στην συνεδρίαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στην Καμπάλα. Τώρα να δούμε τι έγινε με τον, με τον Στολίσκο και την κρίση που ξέσπασε στα νυχτά της Γάζας και αυτά τα τρομερά γεγονότα. Κάτι το οποίο βεβαίως και τράβησε την προσοχή όλων μας. Ο πρόεδρος Μπούζεκ είπε ότι εδώ πέρα πρόκειται για κατάφορη παραβίαση του εθνούς δικαίου και της ε, σύμβασης της Γενέβης. Φυσικά και υπάρχουν αντίθετε φωνέ στο Κοινοβούλιο. Πάντω νομίζω ότι αν ε, προσεγγίσουμε το θέμα απλώ των δικαιωμάτων, αυτό θα είναι ένα βήμα θετικό για την ειρήνευση σε αυτή την πολύπαθη περιοχή. Και σας επαναλαμβάνω ότι με τον πια μόνιμο συνεργάτη μας στο Freedom House θα συζητήσουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι μεταρρυθμίσει στον ελληνικό κόσμο και σα ευχαριστούμε που μα διευκολύνετε ε, κατά την αποστολή στη Washington. Ε, ε, σα προτείνω επομένω στι 23 Ιουνίου σε σχέση με αυτή την πρόσφατη κρίση να συζητήσουμε το, για το τι γίνεται με την κοινωνία των πολιτών στο Ισραήλ. Και κατόπιν εξετάσουμε αυτά τα διφορούμενα ζητήματα όσον αφορά το Ισραηλινό δίκαιο και του κατασταλτικό, του περιοριστικό του χαρακτήρα, να μιλήσουμε με κάποιους ακτιβιστές και φυσικά θα καλέσουμε εκπρόσωπο της πρεσβείας του Ισραήλ. Και όπως σας ε, προείπα θα συνδιοργανωθεί αυτή η εκδήλωση με την ε, αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου για σχέσεις ε, με Παλαιστίνη και Ισραήλ. Επίσης, Είπαμε ότι πήγε στην Κίνα ο πρόεδρος Μπούζεκ και χθε με λεπτομέρειες μου είπε τι έκανε, τι επαφές είχε με ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μου είπε και για τις εκεί δημόσιες δηλώσεις του, αλλά κάτι άλλο θα πρέπει να σας πω, ότι έχουμε τρει, συνάδελφοι, εγώ, η κυρία Όλαν και ο κύριος Μακμίλαν Σκότο, ο αντιπρόεδρος, απευθυνθήκαμε στον πρόεδρο και είπαμε να θίξει τα θέματα των δικαιωμάτων αλλά και τα θέματα του Θιβέτ όταν πάει στην Κίνα. Ξέρετε, εκατοντάδες βρίσκονται φυλακισμένοι. Και τις 10 Μαρτίου 2008 συνελήφθησαν πολλοί στα συλλαλητήρια που γίνανε στη Λάσα, στο Θιβέτ. Πάρα πολλοί και υποφέρουν όλοι αυτοί μόνο και μόνο γιατί προσπάθησαν να ασκήσουν τα θεμελιώδη του δικαιώματα. Επίσης, σε σχέση με την Κίνα, θα πρέπει να σας πω ότι σχεδόν, κατά λάθο συνάντησα τον Ραμπία Καντήρ στην Ουάσινγκτον κατά την αποστολή μα. Και θα θυμάστε ότι είναι η πρόεδρος, η πρόεδρος του Κογκρέσου για το Ουιγκούρ. Not only in Tibet, but also in, in Xinjiang, και συζητήσαμε και για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων στην περιοχή τους. Τη Δευτέρα πήγα στην Ρωσία να υποστηρίξω μια ειρηνική διαδήλωση που έχει σχέση με το άρθρο 31 του Ρωσικού Συντάγματος για το και μου του συναθρίζεστε και αυτό έγινε στην Αγία Πετρούπολη. Ξέρετε ότι μένω πολύ κοντά. 700.000 ε, ήταν αυτοί που συμμετέχουν σε δύο χωριστές ε, διαδηλώσει. Ξέρετε, οι Ρώσοι δεν διστάζουν να εκφράσουν τις απόψει τους να διαδηλώσουν για αυτές και η συμμετοχή μου εκτιμήθηκε πάρα πολύ. ο κύριος Νέμτσοφ ένα από του ηγέτε τη αντιπολίτευση, το είπε δημόσια. Το είπε στον κόσμο ότι η παρουσία μου απέτρεψε την αστυνομία από κατασταλτική άσκηση Δεν ξέρω αν το αμφισβητώ αυτό, αλλά τέλος πάντων ε, ήταν πάρα πολύ τολμηροί, θαραλέοι οι διαδηλωτές. Ε, δεν φοβόντουσαν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο αντιπρόεδρος ε, και και ένας συνάδελφος Ζέμκε και Ντιμ επίσης με βοήθησαν και θα γίνει η επόμενη διαδήλωση τον Ιούλιο, όποιος θέλει που μπορεί να πάει, τέλος πάντων εκφράστε την αλληλεγγύη σα και συμφωνήθηκε στις 31 Μαΐου στις Βρυξέλλες να γίνει επίσης μια διαδήλωση διαμαρτυρία. Επίσης, για τη Ρωσία. Έγινε μια ενημερωτική συνάντηση. Διαβουλεύσεις έψον Ρωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ήταν πιλωτικού χαρακτήρα αυτή η συνάντηση, γιατί για πρώτη φορά η υποεπιτροπή έκανε τέτοιου είδους ενημερωτική συνάντηση με την ε, Επιτροπή την Αρμόδια τη σχέση με την ε, Ρωσία. Εάν θεωρηθεί ότι αυτό το σχήμα βοηθάει, τότε θα το κάνουμε και με άλλες ε, αντιπροσωπείε. Τέλος πάντων αυτό θα το συζητήσουμε αργότερα περαιτέρω. Επίσης, όπως είπαμε, την πρώτη εβδομάδα πήγαμε στην Ουάσιγκτον. Ε, με ενδιαφέρον συναντηθήκαμε με την νέα Αμερικανική κυβέρνηση να ακούσουμε τις απόψεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θεωρήσαμε ότι υπήρξε φιλικό περιβάλλον, φιλική ατμόσφαιρα και επομένω ε, είχαμε με χαρά ε, διαπιστώσει ότι υπάρχουν κοινά σημεία ε, για τον Κουαντάναμο, για την πολιτική των ΗΠΑ όσον αφορά τους κρατουμένους. Είχαμε πει που πάσχει το σύστημα το αμερικανικό σε σχέση με το διεθνές δίκαιο. Και σε σχέση με το κλείσιμο του Γουαντάναμου θεωρήθηκε ότι θα πρέπει να υπάρξει υποστήριξη μέσω αυτών των επαφών. Πάντως, η επιτροπή μας μπορεί να έχει πιο στενή πρακτική συνεργασία με το Κογκρέσο, τον είπα και πιο συγκεκριμένα την αντίστοιχη η Υποεπιτροπή τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Την Επιτροπή των Λάντος. Άρα αυτό το παρακολουθήσουμε το θέμα και τέλος Ιουνίου θα έχουμε την επίσκεψη. Με συνάδελφο της αντιπροσωπείας πάντως ήταν ε, στην Ουγγάντα, στην Καμπάλα μεγάλη την προσωπία που πήγε και έγινε αυτή η συνάντηση για την αναθεώρηση της συνθήκης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, της συνθήκης της Ρώμης. Επίσης έχουμε την συνάντηση του, του τέλους Ιουνίου και όσον αφορά το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σας θυμίζω ότι πρόσφατα περάσαμε κάποιο ψήφισμα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βία στην Ταϊλάνδη. Άλλη ανακοίνωση. Είδατε τι έγινε πρόσφατα με αυτά τα αντικυβερνητικά συλλαλητήρια στην Μπαγκόκ που κατέληξαν στον φόνο τουλάχιστον 85 και τραυματισμό χιλίων ανθρώπων. Επίσης είχαμε ένα σχετικό ε, ψήφισμα και είπαμε ότι θέλουμε μια μερόληπτη ανεξάρτητη επιτροπή να διεξαγαγεί έρευνα για το τι έγινε, ερευνηθούν όλα προς όλες τις πλευρές. Και εμείς ε, τοποθετηθήκαμε σε σχέση με αυτά τα γεγονότα και εκφράσαμε την ανησυχία μας. Σας προείπα ότι η Ταϊλάνδη ήταν από τα θέματα των τριών κατεπηγόντων ψηφισμάτων στην τελευταία ε, συνάντηση τελευταία σύνοδο. Το άλλο ήταν και η Μπούρμα για τις εκλογές που διεξήχθησαν με παντελή έλλειψη δημοκρατικών συνθήκων. Επίσης, κρόσαμε τη δυσαρεσκιά μας σε σχέση με το πώς έχει κατάσταση για τον αποκλεισμό του βασικού δημοκρατικού κόμματος αντιπολίτευση. Το βασικό μας συνομιλητής μέχρι να γίνει πριν από λίγο καιρό η διάσπασή τους ή μπορούμε ήταν το δεύτερο ψήματο και το τρίτο ήταν η θρησκευτική ελευθερία στο Πακιστάν. Αυτό συνέπεσε με την επίσκεψη του Υπουργού Αρμόδιου για τις Μειονότητες στο Κοινοβούλιο. Είχα την χαρά να τον συναντήσω και του είπαμε ότι έχουμε κάποιε επιφυλάξει, ανησυχούμε για δεσμενεί διακρίσει, για τη συμπεριφορά προ τι μειονότητε και κυρίω τι θρησκευτικέ μειονότητε στη χώρα του. Το Δεκοινοβούλιο απευθύνθηκε στην κυβέρνηση και του είπαμε ότι θα πρέπει και η θρησκευτική ταυτότητα και, το θρησκευτικό πιστεύω, το δόγμα που πιστεύουν οι κάτοικοι του Πακιστάν τα πρέπει να φέρνουν ταυτότητα παρά του νόμου κατά τη βλασφημίας. Είναι και τραγικό. Πριν ένα μήνα είχαμε δύο ακτιβιστές των δικαιωμάτων που στην Οαχάκα, ε, στο νότιο Μέξικο, ε, δολοφονήθηκαν Καρίνιο, Μεξικανή και Γιούρι Γιάκολα, μία ή ένας, ένας μάλλον, Φινλανδός. Και συνοδεύαν ένα, ένα κομβό ανθρωπιστικής βοήθειας σε, σε κάποια πόλη στο νότιο Μεξικό, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου έκανε σχετική δήλωση στην Ολομέλεια όταν άρχισε να προεδρεύει. Εγώ έστειλα κάποιες ε, επιστολές και στο Μεξικό θέλουμε να υπάρξουν υπάλληλοι της ΕΕ για ένα άλλο ανθρωπιστικό κομβόι, Καραβάνη που θα φύγει 7η Ιουνίου από το, από το Μέξικο City, την πρωτεύουσα την πόλη του Μεξικού, για τον ίδιο προορισμό και επίσης απευθυνθήκαμε και στις οικογένειες των δολοφονηθέντων. Οι ηθαγενείς εκεί, σε, σε αυτές τις αυτόνομες περιοχές, πρέπει να προστατευτούν. Ε, οι θέσεις τους είναι πάρα πολύ ευάλωτοι. Επίσης, ήρθαμε σε επαφή και με τον Χείρο, τον σύζυγο της ε, δολοφονηθήσης ε, που έπεσαν θύματα αυτών των παραστατητικών που ε, επιτέθηκαν στο καραβάνι το ανθρωπιστικό Βλέπω οι, οι καλεσμένοι μας από την Νόκια και τη Siemens ανυπομονούν. Παρακαλώ υπομονή γιατί λέμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. και θα πρέπει να δούμε το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από μια τέτοια επίθεση στο ανθρωπιστικό κομβολιο Πρώτα πρώτα να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε την ευκαιρία, αυτό το χώρο, το βήμα, ούτως ώστε να έρθουμε και να καταγγείλουμε αυτό το τραγικό γεγονός της 27 Απριλίου μόλις πριν από ένα μήνα που είχαμε αυτό το καραβάνι το ανθρωπιστικό το οποίο επρόκειτο να μεταφέρει κάποια, κάποια, κάποια τρόφιμα στο Σαν Χουάν ε, του της Ουαχάκα όπου έχουμε 800 ε, ηθαγενείς και ε, κάποιοι παραστατιωτικοί που λέγεται Βισόρ επιτέθηκαν και επρόκειτο για ε, για, για ομάδα που χρηματοδοτείται από τον κυβερνήτη της επαρχίας ε, χρηματοδοτείται από τον ορτή στον κυβερνήτη επομένως για να χτυπήσει ε, ε, αυτούς τους ηθαγενείς παρά τη συμφωνία του 69 που υπάρχει που προβλέπει την προστασία τους. Οπότε εμείς είμαστε ακτιβιστέ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα όμως μας κατηγορούν, μας προσάπτουν εγκλήματα, μας διώκουν και πολλοί από εμά ε, δολοφονούνται, υπάρχουν εξαφανίσεις πολλών εξημών και όταν βγαίνουμε δημόσια και καταγγέλουμε όλα αυτά τα οποία γίνονται, που γίνονται σε καθημερινή βάση κατά του λαού της Ουαχάκα. εξήντα δολοφονήθηκαν εκεί, σε αυτό το χωριό, ε, από τον τοπικό κυβερνήτη τον Λουίς Ορτής και πάνω από 500 ε, κρατούνται γιατί ε, διαδήλωσαν για τα δικαιώματά τους. Κανείς δεν κάθισε να διαπιστώσει αν έχουμε διάπραξη εγκλήματος. Και στο χωριό αυτό κάθε μέρα εφίσταται διώξεις ο πληθυσμός γιατί διεκδικεί τα δικαιώματά του, το θεμελιώδη. Η δε κυβέρνηση της χώρας έχει υποχρεωθεί να συνάψει κάποιες ε, διεθνείς συμφωνίες για την προστασία των Ιθαγενών και της κουλτούρας τους. Όμως αυτά όλα μένουν λόγια. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους προσπαθούμε να προστατεύσουμε, υφίστανται επιθέσεις σαν αυτοί που υπέστη αυτό το ανθρωπιστικό καραβάνι. Εμείς ήρθαμε εδώ για να ζητήσουμε την τιμωρία των υπευθύνων αυτού του εγκλήματος, αυτής της ανθρωποκτονίας. Ήδη η κυβέρνηση της χώρας έχει όλα, τα στοιχεία που χρειάζονται ούτως ώστε να προσαγάγει στην δικαιοσύνη τους ε, υπεύθυνους, τους δολοφόνους. Μιλούμε για 800 οικογένειες που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης. Δεν έχουν τα στοιχειώδη, τα βασικά. Δεν έχουν καν φαγητό. Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να υψώσει τη φωνή της και να ζητήσει να ξεκαθαριστεί αυτή η κατάσταση και να ζητήσει τον αφοπλισμό την διάλυση αυτών των προστατευτικών και τη φυλάκιση και την τιμωρία όποιου πρέπει από αυτούς που δρούν στην περιοχή της Οαχάκα. Ήρθε η ώρα η διεθνής κοινότητα να ζητήσει από την κυβέρνηση του Μεξικού να φροντίσει για την πραγματική τήρηση και το σεβασμό αυτών των δικαιωμάτων. Υπεύθυνο είναι ο Ορτής Λουής, ο κυβερνήτης της επαρχίας. Ακολουθεί πολιτική δίωξη αυτών των ανθρώπων. Το μόνο που θέλουν είναι τα δικαιώματα στα συνταγματικά. Το δε βασικό δικαίωμα το οποίο εμείς ζητούμε είναι το δικαίωμα στη ζωή. οι σύζυγος ήταν σε αυτό το καραβάνι. Τη σκοτώσανε. εσείς έχετε την ευκαιρία να απαιτήσετε από την ε, κυβέρνηση να τηρήσετε επεσχημένα σε αυτές τις διεθνείς συμφωνίες. Μπορείτε να τους το ζητήσετε γιατί μόνο μέσω ή μόνο μπορεί να ακουστεί η φωνή μας και να γίνει απονομή δικαιοσύνη. Η Μπέτη Καρίνιο, η γυναίκα μου βέβαια θα ωφεληθεί, έχασε τη ζωή της. Δεν θα ωφεληθεί από την απονομή δικαιοσύνη, αλλά πρόκειται για μια εγκληματική επίθεση και επομένως δεν μπορώ παρά να τα πω αυτά και να σας ζητήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να εκφραστώ. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Όντως πρέπει να γίνει μια ενδελεχής έρευνα για τα εγκλήματα αυτά. Ίσως αυτή η περίπτωση να είναι η ευκαιρία που θέλουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα της ατιμορρησίας που επικρατεί στην Ουαχάκα με διάφορους αντάρτες που εξυπηρετούν τα συμφέροντα της ε, τοπικής ελίτ. Οπότε θα ζητήσουμε, πρέπει να απαιτήσουμε μία ενδελεχή εις βάθους έρευνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα πάμε στην ακρόασή μας για τις νέες ε, τεχνολογίες ε, πληροφορίας και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να δούμε ποια είναι, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που υπάρχουν για τις, από τις νέες αυτές τεχνολογίες, προλαμβάνωμένο και του ίντερνετ, του Twitter, διάφορων άλλων δικτύων, ε, κοινωνικών δικτύων. Είχαμε ξαναπεί ότι θέλουμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό και στην υποεπιτροπή ξεκινήσαμε μια τέτοια συζήτηση με την Σουηδική Προεδρία για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Η υποεπιτροπή λοιπόν αποφάσισε ότι θα πρέπει να γίνει μια μελέτη από την Επιτροπή, από την Κομισιόν. Και κάποιοι από εμά είμαστε και σε επαφή με διάφορες επιχειρήσεις που θα μπορούσαν ίσως να μας, δώσουν κάποιες λύσεις ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των κινδύνων, και πώ μπορούμε να ενισχύσουμε το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω των νέων τεχνολογιών. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Άντριο Κούντεφατ που ε, εκπροσωπεί τους ε, Global Partners και Associates ε, που έκανε την έρευνα δηλαδή για μας έρευνα που έχει τίτλο νέες τεχνολογίες ε, και ανθρώπινα δικαιώματα. Θα του δώσω λοιπόν το λόγο και 10 λεπτά για να μας κάνει την παρουσίασή του. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την ε, δυνατότητα που μας δώσατε και για να κάνουμε την ε, έρευνα και για να σας παρουσιάσουμε τα απορίσματα της σήμερα. Αν μπορούσα να κάνω μια περίληψη, ήταν ότι αυτές οι, είναι οι ε, τεχνολογίες δίνουν τη δυνατότητα να ενισχυθεί η προστασία των δεδομένων σε όλο τον κόσμο, αλλά υπάρχουν ε, φυσικά πολλέ προκλήσει όταν θέλουμε να υποφεληθούμε αυτών των ευκαιριών. Όταν μιλούμε για την ψηφιακή τεχνολογία επί χάρτου, την ε, διαχωρίζουμε σε τέσσερα επίπεδα. Το πρώτο είναι η βασική υποδομή της, της ε, επικοινωνίας, τα τα υλικά δηλαδή, ε, οι συσκευέ κτλ. Α πούμε στην ε, Βρυμανία πριν από κάποια χρόνια στις, ε, διαδηλώσεις ε, η ε, κυβέρνηση έκλεισε όλες τις υποδομές για να μην μπορούν ε, όσοι διαδήλωναν να έχουν επαφή με τον έξω κόσμο. Επίσης διαλειτουργικότητα, σύνδεση με το πώς δηλαδή οι διάφορες συσκευές επικοινωνούν μεταξύ τους. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Όπως ας πούμε η κυβέρνηση του Ιράν χρησιμοποίησε την τεχνολογία των κινητών τηλεφώνων για να βρει ποιοι είναι οι διαδηλωτές που διαδήλωναν εναντίον της κυβέρνησης στις εκλογέ τρίτο επίπεδο επικοινωνίας, οι, εφαρμογε, οι εφαρμογές, οι, ερευνα, οι μηχανές αναζήτησης, εφαρμογές των Windows που, έχουμε, που μας βοηθούν να έχουμε πρόσβαση στη τεχνολογία. Γι' αυτό είναι σημαντικό γιατί οι Κινέζοι ε, επενδύουν πολλή ενέργεια να παρεμβαίνουν ας πούμε, στο ε, επίπεδο αυτό ώστε να μην μπορούν οι πολίτες να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν αυτό το, αυτή τη δυνατότητα για να μην έχουν πρόσβαση σε, ε, σε ευαίσθητο υλικό που δεν θέλουν οι αρχές να το δουν. Και επίσης παρακολούθηση του τι γίνεται, γιατί πολλές φορές σε πολλές ε, χώρες υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει λογοκρισία. Ε, μέσα σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν και το τι θα μπορούσαμε να πούμε πριν από 20 χρόνια, πρέπει να πω ότι λίγοι θα νοιαζόντουσαν πριν από 20 χρόνια για το τι διαβάζει κανεί στις, στις εφημερίδες ή για τις κάμερες που τραβάνε ό,τι βλέπουν στις ειδήσει. Δεν ήταν λοιπόν τόσο σημαντικό αυτό που βλέπαμε κάποτε. Στον σύγχρονο κόσμο όμως αυτά τα επίπεδα, η διαλειτουργικότητα, οι εφαρμογέ το περιεχόμενο, όλα αυτά είναι ε, θεμελιώδος σημασία για να ε, υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον, με όλα αυτά τα επίπεδα, δεν μιλούμε μόνο για ένα εθνικό περιβάλλον το οποίο το ελέγχει η κυβέρνηση. Μιλούμε για ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο εν μέρη το ρυθμίζουν οι διάφοροι κανονισμοί, αλλά το ρυθμίζουν και οι καινοτόμε επιχειρήσει, οι νέε τεχνολογίε και κυρίω οι ίδιοι χρήστε. Γιατί όταν οι χρήστε χρησιμοποιούν την τεχνολογία είναι αυτοί που ακριβώς επαναθέτουν τα όρια αυτού του, αυτού του περιβάλλοντος και θέτουν ε, τις ε, νέες ε, προκλήσεις. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα οικοσύστημα που εξελίσσεται. Δεν είναι ένα ελεγχόμενο σύστημα που ακολουθεί αυστηρού κανόνε, αλλά είναι ένα σύστημα το οποίο, του οποίου τι αξίες πρέπει να επηρεάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Και γι' αυτό είναι πρόκληση αυτή για του φορεί που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί το θέμα δεν είναι απλώ να μιλούμε για τι πολιτικέ που εφαρμόζουμε στα διάφορα αυτά επίπεδα, αλλά είναι και η όλη ε, επεξεργασία τη πολιτική. Πώ δηλαδή μπορούμε να επηρεάσουμε ένα τέτοιο διεθνέ περιβάλλον που το επηρεάζουν τόσο πολλοί διαφορετικοί φορεί, με τόσο, πολύ, με τόσο διαφορετικούς τρόπους. Οπότε το θέμα δεν είναι μόνο τι θέλουμε να κάνουμε, αλλά πώ θα το κάνουμε. Αυτό που αναφέρεται στην ε, έκθεση είναι τέσσερις ε, βασικοί τομείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο πρώτος που είναι στο κεφαλαίο 2 είναι η ελευθερία της έκφρασης. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν ενισχύσει πάρα πολύ τη δυνατότητα που έχουμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας και να συνεργαζόμαστε. Και επίσης τονίζουμε το ότι αυτό δεν είναι απλώ μια διαφορετική τεχνολογία, αλλά ένας διαφορετικός τρόπος επικοινωνίας. Περνούμε, περνούμε σε μια ε, φάση επικοινωνίας από, από ομότιμο σε ομότυπο, Οπότε είναι πιο εύκολη η δημο, ο εκδημοκρατισμός της έκφραση. έκφρασης. Ε, δεν μένει στα χέρια μόνο των ελίτ, της κυβέρνησης, ε, με, μεταφέρεται στην, στα χέρια της κοινωνίας. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για όσους πιστεύουν στην ελευθερία της έκφρασης ως θεμελιώδους ανθρώπινης αξίας. Επίσης, μιλούμε για το ότι υπάρχουν... Ε, πολλά εργαλεία ε, κρυμμένα που περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης. Ξέρουμε ότι το ίντερνετ είναι πάρα πολύ, χρησιμοποιείται πολύ, από εγκληματίες, από τρομοκράτες, από όσους είναι αντίθετοι με τα ανθρώπινα δικαιώματα, από παιδραστές. Ε, υπάρχουν λοιπόν ε, οι ε, πιθανότητες για να χρησιμοποιήσει κανείς ε, το ίντερνετ. Το θέμα είναι να επιβάλλουμε και τους σωστού προορισμού, ώστε να μην καταπατώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και επίσης αναφέρουμε και την περιπλοκότητα αλλά και τι προκλήσεις που έχουμε όταν ε, συνεργαζόμαστε με διάφορους φορείς. Οι πολίτε είναι σημαντικοί παίχτε ό,τι αφορά την ψηφιακή τεχνολογία και σημαντική σύμμαχοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημαντικό ρόλο να παίξει όταν ε, συνεργάζεται με τέτοιου φορεί και με του πολίτε, έτσι ώστε να δούμε πώ μπορούμε να, να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να τα σέβονται όλοι στη δουλειά που κάνει ο καθένα. Εταιρική σχέση μεταξύ ε, περιχειρήσεων και ε, οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπω γίνεται α πούμε στη ΣΥΠΑ. Θέλουμε να υπάρχει συμφωνία από την Κομισιόν ω προς αυτό και πρέπει να δούμε πώ μπορούμε να ενισχύσουμε, να ενθαρρύνουμε τις, ε, τις ε, επιχειρήσεις να επενδύσουν σε τέτοιες νέες ε, τεχνολογίες ε, σεβόμενοι ταυτόχρονα τα, αυτόματα, ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης η ασφάλεια, η εποπτεία είναι πολύ σημαντικέ, γιατί ε, μιλούμε για, το, για τρομοκρατία. Έχουμε δει πολλές φορές ε, χρήση από κυβερνήσεις ε, της ψηφιακής τεχνολογίας για να ενισχύσουν την παρακολούθηση των πολιτών στι ε, στις χώρες τους. Επίσης εξόριξη δεδομένων για να αυξηθεί το μερίδιο της αγοράς η προστασία λοιπόν της ε, ιδιωτικής ζωής των πολιτών χάνει ε, προς όφελος ε, της εκμετάλλευσης της ιδιωτικότητας αυτής από τις εταιρείε. Για το οικονομικό κέρδος δηλαδή και για να μπορεί η κυβέρνηση ίσως να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες. Δεν αρνούμαστε βέβαια ότι οι εταιρείε χρειάζονται τέτοιες προσωπικές πληροφορίες, τέτοια δεδομένα, ούτε ότι η κυβέρνηση μπορεί να τα χρειαστεί κάποια στιγμή για να αντιμετωπίσει θέματα τρομοκρατικών απειλών. Αλλά υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη να παρουσιαστούν αποδείξεις που θα έδιναν λόγο, που θα έδιναν λόγο στις κυβερνήσεις να περιορίσουν την ελεύθερη έκφραση των, των πολιτών τους. Να δούμε δηλαδή ποιοι είναι αυτοί οι κίνδυνοι, ποιε είναι αυτές οι που υπάρχουν και που, που επιβάλλουν τον περιορισμό αυτό στους πολίτες. Τρίτο, στο κεφάλαιο 4, Τονίζουμε τη σημασία των ωφελών της ψηφιακής τεχνολογίας για την επιστημονική πρόοδο και την πρόσβαση στην εκπαίδευση. Πιστεύουμε ότι αυτές οι τεχνολογίες έχουν, έχουν δημιουργήσει ένα εξαιρετικό δυναμικό για την εκπαίδευση. Παρ' όλα αυτά αυτό έχει, να κάνει, έχει πάρα πολλούς κινδύνους για τον τομέα της, των ε, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα οποία ε, χρησιμοποιούν ε, τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις χωρίς να δίνεται όμως καμία σημασία στα ε, πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. Γι' αυτό δημιουργούνται τώρα νέοι πιο αυστηροί α, κανόνες για τα πνευματικά δικαιώματα και αυτό αναφέρεται στο κεφάλαιο 4. Τελευταίο, η κεφάλαια 5 και 6. Μιλούμε για την σημασία της ανάπτυξης, της ισότητας, Τονίζουμε ότι με την, με την επιφύλαξη των περιορισμών υπάρχει ε, ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών και στις πιο αναπτυσσόμενες χώρες. Υπάρχει λοιπόν μεγάλο περιθώριο να ενισχύσουμε πιο το, την ε, ανάπτυξη των ε, τεχνολογιών αυτών και στις, στην Ήπεθρο. Επίση οι μειονότητες πρέπει να έχουν πρόσβαση στις τεχνολογίες αυτές, οι άνθρωποι με αναπηρία πρέπει να έχουν ε, πρόσβαση στις ψηφιακές ε, τεχνολογίες και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό πρέπει να το ε, ενισχύσει. Επίσης, στο κεφάλαιο 7 λέμε ποιος θα είναι ο ρόλος που πρέπει να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην, στην όλη πολιτική για τις ψηφιακές τεχνολογίες. οι εσωτερικέ πολιτικέ, ε, που είναι βέβαια θέμα κυρίω τη της ε, Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, έχουν, μια σημαντική, έχουν σημαντικές συνέπειες στο πώ καταλαβαίνουν οι υπόλοιποι και πώ εφαρμόζουν τι ε, αξίε τη Ένωση, α πούμε έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό για να δούμε πώς μπορούμε να επηρεάσουμε τα πράγματα παγκοσμίω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, ε, ειδικά σε ό,τι αφορά την προώθηση ε, των τεχνολογιών για την διακυβέρνηση από τον ΠΟΕ, από τον Οργανισμό για την ε, Πνευματική Ιδιοκτησία και μέσω πολυμερών ε, συμφωνιών σε τέτοιου είδους ε, εμπόριο για, το, για τα διπλώματα βρεσιτεχνίας. Και το πνευματικά... Μπορεί να χρησιμοποιήσει φυσικά και τις διπλωματικές της ικανότητες έτσι ώστε να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα στον ψηφιακό κόσμο. Υπάρχουν δυνατότητε εταιρική σχέσης με τις Ηνωμένε Πολιτείε, με τη νέα Αμερικανική κυβέρνηση και μετά από την ομιλία του Προέδρου τον Ιανουάριο και την ομιλία του Καρλ Μπίλτ πρόσφατα. Είχαμε συζητήσεις για την προετοιμασία του εγγράφου αυτού με ανώτερους υπαλλήλους του State Department υπογραμμίσαμε την επιθυμία του Στέντι Πάρκμαν να συνάψει στενές σχέσεις με Ευρωπαίους πολιτικούς για να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα στον υπόλοιπο κόσμο. Έχουμε δηλαδή αρκετέ δυνατότητε για μια ουσιαστική μορφή συντονισμού ανάμεσα στι κυβερνήσει μα Και τέταρτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εργαστεί με κυβερνήσει, με την κοινωνία των πολιτών, με μη κυβερνητικέ οργανώσει, έτσι ώστε να βελτιώσει τα επιχειρηματικά πρότυπα και τι καθημερινέ πρακτικέ που θα διευκολύνουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέλο έχουμε κάποιε συγκεκριμένε συστάσει τι οποίε θα θέλαμε να κάνουμε προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον, να υιοθετήσει ε, σε περιπτώσεις κρίσης σε επικοδομητικά διπλωματικά μέτρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να υπογραμμίζεται σε όλες τις μορφές διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο σεβασμός online των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να χαρακτηρίζει και τις εμπορικές διαπραγματεύσεις και θα πρέπει να είναι θέμα το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται σε συζητήσεις και με τα Ηνωμένα Έθνη και με όλους τους θεσμούς οι οποίοι συνδέονται με εθνικές κυβερνήσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί κυρίως στις επαφές που έχουμε με τις Ηνωμένε Πολιτείες και την Βραζιλία. Υπάρχει ανάγκη επίσης έτσι ώστε να υπάρξουν περαιτέρω έρευνες για να επιληθούν προβλήματα περίπλοκα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι αποφάσεις που θα πρέπει να λαμβάνονται να βασίζονται σε αποδείξεις και σε τεκμήρια και όχι σε προκαταλήψεις και σε φοβία. Θα πρέπει επίσης να πάρουμε μέτρα με όλους τους τρόπους έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν όσο καλύτερα γίνονται οι τεχνολογίες οι οποίες είναι διαθέσιμες. Θα πρέπει επίσης να βελτιώσουμε την ικανότητα των εμπλεκομένων εταίρων να επιλύουν τα προβλήματα, να λειτουργούν προληπτικά και σε επίπεδο επιχειρήσεων και κυβερνήσεων και να προωθούν την καινοτομία και τις ετορικές σχέσεις για να βελτιώσουν ακριβώς την καινοτομία. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ την προώθηση και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα φέρει σε επαφή την κοινωνία των πολιτών με τους ειδικού στα ηλεκτρονικά για να γνωρίσουμε τις δυνατότητες που μας παρέχουν να προχωρήσουμε και στη δημιουργία μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις επικοινωνίες, να αναπτύξουμε ίσως και κάποια κέντρα ε, βέλτιστων πρακτικών για την χρήση των νέων ηλεκτρονικών μέσων και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων online. Υπάρχουν κάποια προβλήματα, υπάρχουν κίνδυνοι, οι εχθροί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες με αποτελεσματικό τρόπο, κινητοποιούνται και θα πρέπει και το κίνημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τη δική σας υποστήριξη να κινητοποιηθεί και αυτό με τη σειρά του. Ευχαριστώ τον κύριο Πούντενφατ. Uh, θα επανέλθουμε στις συστάσεις σας κύριε Πούντενφατ. Νομίζω ότι θα τη σχολιάσουν και οι υπόλοιποι ομιλητές. Έχω τη χαρά τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Φασίσκο Σίσα Βάγνερ, εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα θέματα του ελέγχου του διαδικτύου. Κύριε Σίσα Βάγνερ, πείτε μας τη γνώμη σας για το διαδίκτυο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα. Να πούμε για αυτή την έκθεση που χθε εγκρίθηκε στην Επιτροπή Βιομηχανία και Ενέργεια να το εντάξουμε σε, ένα πλαίσιο τόσο να καταλάβει ο κόσμο που πρόκειται. Έγινε αυτή η Επιτροπή, όπω θυμάστε, στα, στα, πλαίσια τη δουλειά τη Επιτροπή ε, Έρευνα Βιομηχανία και Ενέργεια. Και ε, ήταν σε συνέχεια μια ε, ανακοίνωση που εξεδόθη από την ε, Επιτροπή. Διακυβέρνηση του διαδικτύου. Τα επόμενα βήματα. Αυτό ήταν ο τίτλος. Και το βασικό μέλημα της ε, Κομισιόν όταν μας διαβίβασαν αυτή την ανακοίνωση για τις ανησυχίες τους για τη διακυβέρνηση του ίντερνετ αφορούσε τον ρόλο μιας Αμερικανικής οργάνωσης που διέπεται από το δίκαιο της πολιτείας Καλιφόρνιας τι μπορεί να κάνει δρώντας σε όλο τον κόσμο μέσω του ίντερνετ δηλαδή αυτά τα domain name αυτές οι διευθύνσεις του ίντερνετ ε, ρυθμίζονται από μία εταιρεία ιδιωτικού δικαίου, ε, από ένα δημόσιο πρόσωπο, από, συγγνώμη, από ένα νομικό πρόσωπο ε, ιδιωτικού δικαίου, το οποίο δεν διέπεται καν από το Ομοσπονδιακό Αμερικανικό Δίκαιο, αλλά από το δίκαιο μια εκ των πολιτιών, τον είπα. Και αυτοί επομένω δίνουν, αυτοί μοιράζουν, αυτοί, αυτοί διαχειρίζονται όλε αυτέ τι διευθύνσει του Ιντερνετ, αυτά τα domain name για, όλο τον κόσμο, για όλο τον το πλανήτη. Οπότε, το, το μέλημα όλων των Ευρωπαίων τη της Κομισιόν συγκεκριμένα ήταν ότι για μας είναι κάπως παράδοξο, είναι περίεργο ένα, μια τέτοια εταιρεία, κάποιος ιδιώτης να, να, να έχει τέτοια δικαιώματα. Πάντως, όσο πράξουν και να φαινόταν, η Κομισιόν σε καμία στιγμή δεν πρότεινε να μεταβληθεί η κατάσταση. Σε καμία στιγμή. Και ακολούθησε την πεπατημένη για, για όλες τις συζητήσεις για το Ιντερνετ. Έχουμε αυτό το φόρμα τη στο του Ιντερνετ και το πρόβλημα αυτό εκεί έχει αναγύψει πολλές φορές. Οπότε ουδέποτε κανένας, κανένας από τους εκεί ε, εκπροσώπους του καθενός δεν εκφράστηκε μια τέτοια πρόθεση μεταβολής. Καμία εναλλακτική δεν προτάθηκε σε σχέση με ε, αυτόν τον οργανισμό που είπαμε, που είπαμε ότι είναι ιδιωτικού δικαίου και βέβαια έχει κάποια σχέση με την κυβέρνηση των ΗΠΑ και υπάρχει κάποια μόργη σύμβαση που του συνδέει με την κυβέρνηση, η οποία κυβέρνηση εποπτεύει την οργάνωση αυτή. Έτσι έχει η κατάσταση και αυτά μας εξηγεί στο κείμενο της Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μας ρωτάει τι πρεσβεύουμε ως κοινοβούλιο για το πρόβλημα. Πάντως, η Κομισιόν δεν θεωρεί ότι η κατάσταση έχει κακό, γιατί όσο και να είναι παράδοξο πλευρά νομική, τουλάχιστον για τη δική μας τελείωση των πραγμάτων, παρόλα αυτά το σύστημα αποδίδει, λειτουργεί. Άρα, αφού λειτουργεί, δεν το πειράζουμε. Αυτό βέβαια που μα απασχολεί είναι αν υπάρχει διαφάνεια σε αυτήν την οργάνωση, ε, σε ποιον είναι υπόλογη ε, αυτή η οργάνωση, τι γίνεται, πώς είναι να έχουμε όσο γίνεται περισσότερη εκπροσώπηση ε, περισσότερων κρατών. Άρα θα πρέπει να γίνει κάποιος εκδημοκρατισμός αυτού του οργανισμού. Να υπόκειται σε κάποιο έλεγχο, να είναι κάπου υπόλογος αυτός ο οργανισμός. Όλα αυτά τα διατυπώνουμε στην εκθέση αυτή, η οποία συνετάγει στα πλαίσια των εργασιών τη Επιτροπή Βιομηχανία. Αυτό ήταν επομένω το βασικό πρόβλημα. Τώρα. Όπως ακριβώς είπε και ο προλαλή σα, ήταν άρτια αυτή η έκθεση και σήμερα στο ίντερνετ εμφανίζονται όλα τα θέματα για όλο τον κόσμο. Και βέβαια δεν μπορούσαμε παρά να μην ε, θίξουμε στο κείμενό μας το θέμα της άσκησης των θεμελιωδών ελευθεριών. Γιατί και, στο, και το Ιντερνετ είναι χώρος όπου πρέπει κανείς να μπορεί να ασκήσει τα βασικά του δικαιώματα, ας πούμε την ελευθερία της, το δικαίωμα στην, στην έκφραση της γνώμης Το Οπότε έχουμε εδώ πέρα αυτό το νομικό πρόβλημα και αυτό το πράγμα που πηγάζει από αυτή την, την ιδιότυπη, τη μοναδική σε όλο τον κόσμο οργάνωση, οργανισμό μας δόθηκε η ευκαιρία επομένως να μπορέσουμε να προβούμε σε κάποιες διευκρινήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διαδίκτυο. Αφετηρία μας ήταν ότι το διαδίκτυο είναι παγκόσμιο αγαθό και δημόσιο. Οπότε και εμείς είπαμε ότι αντίστοιχα θα πρέπει η διαχείριση να γίνεται με συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ετάχνουμε δε υπέρ τη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όπω αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα διατυπώνονται από τι συνθήκε που διαβούν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το διαδίκτυο. Σα πρέπει τώρα στην τρίτη παράγραφο του κειμένου που λέει ότι οι αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώ όπω αναγνωρίζουν και διατυπώνονται από την συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι θεμελιώδει αξίε και είναι στόχοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την πολιτική τη για την κυβέρνηση του διαδικτύου. Απευθύνει δέκληση στη θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στα κράτη-μέλη για να προστατεύσουν αυτέ τι θεμελιώδει αξίε σε όλα τα διεθνή φόρα και συγκεκριμένα σε εκείνα όπου συμμετέχουν χώρε οι οποίε δεν συμμερίζονται γενικώ επί τις αξίες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά λέει αυτή η έκθεση που είχα την τιμή να συντάξω για την κοινωνική μα επιτροπή. Απίθυνο λοιπόν έκκληση για την πρόσπιση αυτών των ελευθεριών σε όλα τα διεθνή φόρα. Όλα τα οποία ασχολούνται με το Ιντερνετ, α πούμε, το, το φόρουμ για τη διακυβέρνηση Ιντερνετ, αλλά και υπάρχουν και άλλα. Και ιδίω τονίζουμε το γεγονό ότι υπάρχουν κάποιε χώρε που δεν συμμερίζονται αυτές τις ευρωπαϊκές πούμε αξίες και ελευθερίες. Επομένως, σε σχέση με αυτές τις χώρες θα πρέπει εμείς να αντιτάξουμε αυτές μας τις, ε, τις ιδέες, τις αξίες που κατοχυρώνονται με την ε, συνταγματική συνθήκη μας. Οπότε, σε σχέση με αυτή την πολιτική που θα πρέπει να ασκήσουμε, είπαμε στην 8η παράγραφο τη έκθεση ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, θα πρέπει να υπάρχει πολυμερής, πολυμερής σχέση και δομή και θα πρέπει να τηρούν και τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, όπως ορίζουν το κοινοτικό δίκαιο και οι θεμελιώδεις ε, ελευθερίες. Οπότε θέλουμε να είναι ανοιχτό το διαδίκτυο και είπαμε ότι θέλουμε κατηγορηματικά να καταδικάσουμε τους περιορισμούς προσβασιμότητας στο ίντερνετ και κάποιο είδους ε, φίλτρα, μπλοκαρίσματα, λογοκρισία και όποτε υπάρχει κάποιο είδους επιβολή περιορισμού της προσβασιμότητας στο ίντερνετ αν κρυθεί αναγκαία ας πούμε όταν ε, έχουμε ε, κάποιες δικαστικές ανακριτικές πράξεις κατά κάποιων εγκλημάτων όπως με παιδική πορνογραφία θα πρέπει οι περιορισμοί αυτοί να γίνονται όπως ορίζεται από τον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και όπως ορίζει η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου για τα θεμελιωδικαιώματα. δικαιώματα. Αυτό το πνεύμα διαπνέει το κείμενό μας και εκμεληθήκαμε την ευκαιρία που μας δόθηκε για να αποφανθούμε όσον αφορά αυτόν τον θεμελιό, αυτόν τον οργανισμό και με την ευκαιρία αυτή που είπαμε όλα αυτά το επιτεθούμε τόσο σημαντικά. Και είπαμε ότι απευθύνουμε έγκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτως ώστε να υπάρξει συντονισμός όλων των πολιτικών που σχετίζονται με το ίντερνετ. Θεωρούμε ότι αυτό είναι σημαντικό. Πολύ πολύ επιμείναμε πάνω σε αυτό. ευρωπαϊκή πολιτική που θα πρέπει να είναι ομοιογενής και συνεπής. Να ακούγεται η φωνή της Ευρώπης μία. Και αυτή η μία και μοναδική φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην να, ε, γίνεται για να αποφύγουμε την, την πολυφωνία, την κακοφωνία των 27 διαφορετικών χωρών που είναι μέσα. Αλλά είπαμε να μην το ξεχνάμε. Δεν θα πρέπει να υπάρχει διαφωνία μεταξύ των δεσμικών οργάνων του Συμβουλίου, Κομισιών και Κοινοβουλίου. Αυτή είναι η έκκληση που απευθύνομαι. Ούτω ώστε να σταματήσουν όλε αυτές οι δυσλειτουργίε, οι αντιφάσεις και έτσι ξεκάθαρη και ενιαία να ακούγεται παντού για τον τερνετή φωνή της Ευρώπης και έτσι να γίνεται η προστασία, η προώθηση αυτών όλων των βασικών μας αξιών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σώσα Βάγναρ. Η παρουσία σας στην υποεπιτροπή μας είναι ένα καλό παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας τις εργασίες άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Λουσί Μωριγιό, εξ ονόματος των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαστε μια διεθνής οργάνωση η οποία υπερασπίζεται το δικαίωμα του να ενημερώνει κανείς και να ενημερώνεται. where the mainstream media is under the control of the regime, we've seen that bloggers, cyber dissidents, Thank you. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε λοιπόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη Βυρμανία και σε άλλες χώρες και το διαδίκτυο έχει γίνει ένα νέο μέσο και για τους προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε χώρες όπως το Βιετνάμ, η Λευκορωσία, η Κούβα και άλλες. Ο τίτλος της έκθεσης που κάνουμε έχει σαν υπότιτλο μάλλον η έκθεση την οποία προετοιμάζουμε «Εχθροί στο Ιντερνετ». Ένα από τα ευρήματα της έκθεσης αυτής είναι ότι οι χώρες οι οποίες επηρεάζονται από διάφορες μορφές λογοκρισίας έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Και είμαστε γύρω στις 60 χώρες, κάτι το οποίο είναι θα έλεγα μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Η λογοκρισία στο ίντερνετ είναι μια προτεραιότητα για ορισμένα καθεστώτα αλλά υπάρχουν ε, κάποια εθνικά διαδίκτυα τα οποία είναι ανεξάρτητα από το παγκόσμιο διαδίκτυο, τον παγκόσμιο ιστό όπως τον γνωρίζουμε εμείς. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διώξεις. 120 άνθρωποι που εκφράστηκαν ελεύθερα στο ίντερνετ είναι σήμερα φυλακισμένοι σε διάφορα μέρη του κόσμου. Από τη μία βλέπουμε τον αυξανόμενο έλεγχο αυτών των κυβερνήσεων και από την άλλη βλέπουμε την επιθυμία των πολιτών να αντισταθούν στη συγκεκριμένη αυτή πίεση. Η, θα έλεγα το αποτέλεσμα του αγώνα ανάμεσα στους ανεξάρτητους πολίτες του διαδικτύου από τη μία και στα κατασταλτικά καθεστώτα από την άλλη ε, θα, έλεγα η κατάληξη θα κρυθεί από τα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε διάφορα επίπεδα μεταξύ των οποίων και στο τεχνολογικό επίπεδο. Κάποιες από τις ε, κυβερνήσεις προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν σαν μέσο ελέγχου τις ίδιες τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στο διαδίκτυο. Οι εταιρείες αυτές βρίσκονται σε αρκετά δύσκολη κατάσταση. Πολλοί πίστευαν ότι ο πρώτος λογοκριτής στην ουσία ήταν ε, η Κίνα βέβαια και η παρέμβασή της δεν μπορούσε να αγνοηθεί. Και παρά τις εκκλήσεις για περισσότερη παρουσία στις χώρες αυτές, οι εταιρείε ένιωθαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν κάποια σημαντικά πράγματα. Η Microsoft, η Yahoo, η Google δεν ε, αντιστάθηκαν καθόλου ουσιαστικά και μάλιστα η Yahoo προχώρησε και στην καταγγελία ορισμένων συγκεκριμένων δημοσιογράφων οι οποίοι μάλιστα συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν και έχουν καταδικαστεί σε 10 χρόνια φυλάκιση. Τώρα η Google αποφάσισε να σταματήσει τη λειτουργία της μηχανής έρευνάς της ε, στα κινέζικα και στρέφει τους ε, χρήστες της στη μηχανή έρευνας της Google στο Hong Kong ε, η οποία ε, ναι μεν είναι προσβάσιμη στους κάτοικους της υπηρετικής Κίνας αλλά μόνο με περιορισμένο κινέζικο λεξιλόγιο. Εν πάση περιπτώσει τώρα υπάρχει μια γνωστοποίηση γενικότερη σε σχέση με, το, με τη μέθοδο που ακολουθείται για την καταστολή και ο κόσμος έχει αρχίσει να αναρωτιέται τι είναι αυτό το οποίο προσπαθεί να τους αποκρύψει και από τι προσπαθεί να τους απομονώσει η κινέζικη κυβέρνηση. Μια άλλη υπηρεσία του διαδικτύου, η Good Andy, αποφάσισαν ότι δεν θα πολλούν ε, κινέζικα, κινέζικους ιστοτόπους ε, γιατί θεωρούν ότι δεν μπορούν να ελέγξουν από εκεί και πέρα το μέγεθος της καταστολής. Υπάρχει η εκστρατεία εναντίον της πορνογραφίας στην Κίνα, η οποία φύγει αυτούς που δεν πρέπει. Έχουν επιβληθεί σκληρότατες καταδίκες σε δημοκράτες και σε ανθρώπους που υπερασπίζονται την ελεύθερη έκφραση στο διαδίκτυο. και αν θέλει κανείς να ανοίξει μια ιστοσελίδα στην Κίνα, ένα ιστότοπο μάλλον στην Κίνα, πρέπει να παρουσιαστεί ο ίδιος προσωπικά και αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πια η ανωνυμία online που ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά θα έλεγα του διαδικτύου και τώρα καλούνται οι χρήστες να ανακοινώνουν το όνομά τους. Λοιπόν, υπάρχει μια σοβαρή πίεση και προς τις ξένες επιχειρήσεις οι οποίες προσπαθούν να παρέχουν πληροφορίες στους Κινέζους Νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να ακολουθηθούν ορισμένες επιχειρηματικές αποφάσεις οι οποίες ε, θα λάβουν υπόψη τους το ότι τα προϊόντα τα οποία παρέχουν δεν διατίθενται στα πλαίσια ενός ελευθέρου διαδικτύου. Δεν ισχύει στην περίπτωση της Κίνας σαν παράδειγμα ένα ελεύθερο, απελευθερωμένο και προσβάσιμο σε όλους διαδίκτυο. Άλλες επιχειρήσεις όπως η Microsoft και η Google δεν θέλουν να αλλάξουν ε, τις πολιτικές τους. Η Microsoft μάλιστα υποτιμά συστηματικά τη σημασία της λογοκρισίας στην Κίνα. Νομίζω ότι χάνει μια ευκαιρία ή χάνουμε όλοι μια ευκαιρία να έχουμε ενιαίο μέτωπο απέναντι στις κινέζικες πρακτικές. Αυτά όλα ισχύουν φυσικά όχι μόνο για τις εταιρείες στο διαδίκτυο αλλά και για τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες στο διαδίκτυο γιατί εκατομμύρια εκατομμυρίων άνθρωποι ε, χρησιμοποιούν ε, το διαδίκτυο μέσω των μικρών φορητών τηλεφώνων τους. Υπάρχουν ιταλικές εταιρείες οι οποίες έχουν, είναι ιδιοκτήτριες άλλων εταιριών στην Άπο Ανατολή, στην Κίνα, στο Βιετνάμ Υπάρχει επίσης ε, γερμανικές επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν φάσματα ε, ε, επικοινωνιών σε χώρες όπως η Βόρεια Κίνα, η Βόρεια Κορέα, συγγνώμη, και γενικότερα υπάρχουν εξελίξεις στις σχέσεις ανάμεσα στις επιχειρήσεις του τομέα και στις διάφορες χώρες. Και θα ακούσουμε με προσοχή και τους εκπροσώπους της Nokia Siemens για το ότι τα δίκτυά τους υφίστανται περιορισμούς σε σχέση με ορισμένες χώρες ε, στο Ιράν γιατί η Nokia Siemens πολλούν υλικό ηλεκτρονικό στο Ιράν και μεταφέρουν πληροφορίες εις βάρος των αντιστασιακών της χώρας αυτής κάτι το οποίο η Nokia μέχρι τώρα το αρνείται. Θα ακούσουμε τις απόψεις που έχετε γύρω από αυτό. Λοιπόν, οι τεχνολογίες ενημέρωσης και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα έλεγα είναι ιδιαίτερα διασυνδεδεμένες μεταξύ τους. Ε, υπάρχει θα έλεγα μια σωστή συνεργασία με τις περισσότερες χώρες και τους μηχανισμούς που ελέγχουν την κυκλοφορία των ιδεών και των πληροφοριών στο διαδίκτυο και θα τελειώσω με ορισμένες συστάσεις, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει, όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής. Θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι, οι εταιρείε στον τομέα της ηλεκτρονικής να μπορέσουν και να καταλήξουν σε ένα κώδικα συμπεριφοράς για τη λειτουργία τους σε λιγότερο ελεύθερες χώρες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό για μας. Δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτό αρκεί. Θα θέλαμε να υπάρξουν κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις έτσι ώστε αυτό θα πρέπει να γίνεται χωρίς να φέρνουμε αντιμέτωπους τις εταιρείε και τις κυβερνήσεις που θέλουν να καταστήλουν την έκφραση μέσα από το διαδίκτυο. Το Αμερικανικό Κογκρέσο υιοθέτησε ένα νόμο που έχει σαν στόχο να αποτρέψει τις επιχειρήσεις να συνεργαστούν με λογοκριτές σε διάφορες χώρες. Θα θέλαμε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει προς την κατεύθυνση αυτή. Προτάθηκε και μία οδηγία την οποία είχε προτείνει ο Μάτενς ε, το 2008 στο προηγούμενο κοινοβούλιο και θα θέλαμε να δούμε τι θα γίνει με την πρόταση για τη συγκεκριμένη οδηγία. Θα θέλαμε περισσότεροι βουλευτές να υποστηρίξουν ένα τόσο σημαντικό κείμενο. Όλες οι ρυθμίσεις θα πρέπει να ζητούν από τις επιχειρήσεις να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από τις επιχειρηματικές τους πρακτικές. Θέλουμε οι επιχειρήσεις αυτές να ανθίστανται στα αιτήματα των κρατικών μηχανισμών ε, τα οποία απαιτούν λογοκρισία. Καλούνται οι εταιρείες αυτές ε, να υπόκεινται φυσικά στους τοπικούς νόμους και ίσως ε, αυτό να ε, οδηγεί σε λύσεις όπως σαν παράδειγμα οι εταιρείε αυτές να μην εγκαθίστανται σε χώρες όπου υπάρχει λογοκρισία αλλά σε χώρες άλλες πιο ελεύθερες. Ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι να υπάρξει έλεγχος στην εξαγωγή ε, υλικού, hardware και ε, software που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους κυβερνήσεις έτσι ώστε να συλλέγουν ελευθερίες εις βάρος των δημοκρατικών στοιχείων στις χώρες τους. Η, Ευρωπαϊ... η κοινοτική ευρωπαϊκή πολιτική και οι διπλωμάτες της Ένωσης θα πρέπει να πιέζουν όλο και περισσότερο για την κατάργηση της ε, λογοκρισίας online και επίσης ε, να υπερασπίζονται αυτούς οι οποίοι ανθίστανται μέσω του διαδικτύου. Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και στα πλαίσια των εμπορικών συμφωνιών και θα πρέπει τα στόπινα δικαιώματα να ε, γίνονται αντικείμενο εξέτασης αν υπάρχει σεβασμός τους και online. see also the European Union encourage efforts to help dissidents secure their communication, you know, help all these proxy initiatives, tools to get around censorship. We believe it's a critical moment to protect human rights online and this means encouraging Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε λοιπόν τις επιχειρήσεις να, σεβε... να σέβονται όλο και περισσότερο την ελεύθερη έκφραση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μωριό. Certainly Ας προσπαθήσουμε τώρα να δούμε πώς όλα αυτά φαίνονται από πλευράς των ιδίων των επιχειρήσεων. Με μεγάλη χαρά βλέπω ότι έχουμε εδώ εκπροσώπους της Google και του δικτύου Nokia Siemens. και εκπροσώπους επίσης ε, της ε, κινέζικης επιχείρησης Dynasty TV. Ας προσπαθήσουμε να δούμε λοιπόν πώς οι επιχειρήσεις ε, βλέπουν τα πράγματα τα οποία εξέτασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαν παράδειγμα στο Ιράν για τις διώξεις και την καταστολή της κοινωνίας των πολιτών. και πώς διώχθηκαν ακριβώς μέσω της χρήσης κινητών τηλεφώνων κτλ. Λοιπόν, ο εκπρόσωπος της Nokia Siemens Network θα πάρει το λόγο. Ελπίζω να έχουμε αρκετό χρόνο, γι' αυτό παρακαλώ αν μπορείτε να μιλήσετε γύρω στα 8 λεπτά για να μπορέσει να γίνει και συζήτηση μετά. Μην μιλάτε ιδιαίτερα γρήγορα βέβαια. Αν χρειάζεται πάρτε ένα-δύο λεπτά περισσότερο για να γίνετε κατανοητός όχι όπως η προηγούμενη κυρία. Είναι υπεύθυνο για θέματα επιχειρήσεων και marketing στην Nokia Siemens. Θα μας μιλήσει για τις... Now very much linked with the European Parliament's resolution on, on January. So, Mr. Friends, welcome and please take the floor. Great. Well, thank you very much. Για τον έλεγχο των τηλεπικοινωνιών μέσω κινητών τηλεφώνων. Είναι δύσκολο να μιλήσω 8 λεπτά και να μιλήσω και αργά κιόλα. Γι' αυτό θα μου πείτε ακριβώς πώς θα πρέπει να το κάνω. Εν πάση περιπτώσει, εγώ εξετίμησα τα σχόλια που έκαναν οι προηγούμενοι ομιλητές όταν είπατε ότι οι εταιρείε αντιμετωπίζουν δυσκολίες και βρίσκονται σε δύσκολη θέση, αυτό είναι αλήθεια. Πράγματι, πολλές φορές αντιμετωπίζουμε δυσκολίες και χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων εσάς έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μέσα σε ένα περιβάλλον που αλλάζει συνεχώς. μπορούμε να προχωρήσουμε και σε ανεπίσημες επαφές ε, ε, με σας και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε πιο συχνά στο μέλλον. Λοιπόν, μου ζητήθηκε να μιλήσω σήμερα για τις εμπειρίες των δικτύων Nokia Siemens σε σχέση με το Ιράν και τη χρήση των, της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών στη χώρα αυτή για την καταστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα το κάνω αυτό, θα μιλήσω όμως και για κάποια ευρύτερα θέματα και για κάποια από τα μαθήματα που πήραμε από τις εμπειρίες αυτές. Πρώτον, η εμπειρία μας σε σχέση με το Ιράν. Το 2009 οι ειδήσει αναφέρθηκαν στην παράδοση τεχνολογιών ελέγχου από την Όκια στο Ιράν δώσαμε βάση περιπτώσει συστήματα δικτυακά για τις δύο μεγάλες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας του Ιράν καλύπτουμε με τα μηχανήματά μας το 1 τρίτο των δικτύων και επίσης τους δώσαμε και δυνατότητες και στις δύο εταιρείες έτσι ώστε να παρακολουθούν κάποιες τηλεφωνικές ε, ε, συνδιαλέξεις. Οι μέθοδοι γενικά παρακολούθησης των συνδιαλέξεων είναι οι δυνατότητες οι τεχνικές που έχουν οι δημόσιες αρχές να ελέγχουν τις τηλεπικοινωνίες. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει και στο, ε, συντακτικό, στο συνταγματικό χάρτη, αν θέλετε, της Διεθνούς Τηλεπικοινωνιακής Ένωσης και ακολουθεί συγκεκριμένα επίσημα standards όπως τα έχει ορίσει το Τηλεπικοινωνιακό Διεθνές Ινστιτούτο όλες οι χώρες ζητούν από τις εταιρείες της κινητής τηλεφωνίας να έχουν τέτοια συστήματα ελέγχου. Και γι' αυτό υπάρχουν σε όλα τα συστήματα τα οποία λειτουργούν στον κόσμο, ακόμα και σε αυτά που χρησιμοποιείτε εσείς εδώ σήμερα. Και αυτό γίνεται για πολύ σωστούς λόγους, για την καταπολέμηση ας πούμε παιδικής τρομογραφίας, πορνογραφίας, συγγνώμη, της τρομοκρατίας και επίσης ε, ε, καταπολέμησης της εμπορίας ναρκωτικών. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για το ποιος είναι αυτός ο οποίος παρακολουθεί τις συνδιαλέξεις και για το ποιος θα πάρει τις πληροφορίες που θα προέλθουν από τις παρακολουθήσεις αυτών των τηλεφώνων, τις υποκλοπές αν θέλετε. Έτσι θα μπορέσουμε, έτσι γίνεται συνήθως, παίρνουν οδηγίες και διαταγές από τις αρμόδιες αρχές, ακολουθούνται ε, θα έλεγα όλες οι μέθοδοι ε, έτσι ώστε να είναι νόμιμες. Βέβαια και τα ενεργά και τα παθητικά στοιχεία του συστήματος υποκλοπών θα πρέπει να είναι πλήρως αναγνωρισμένα από την Διεθνή Τηλεπικοινωνιακή Ένωση μετα... και έτσι όλες οι χώρες έχουν την δυνατότητα να προχωρούν σε υποκλοπές. Οι δύο αυτές τεχνολογίες όμως αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο από την επιχείρησή μας. Εμείς εξηγούμε τη διαφορά που αντιμετωπίζουμε αυτές τις δύο τεχνολογίες και από τεχνικές διαφορές μεταξύ τους και από τους κινδύνους σε, ανθρώπινα, σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εμείς βασικά συνεργαζόμαστε με εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, παρέχουμε υπηρεσίες. Το παθητικό στοιχείο είναι κάτι στο οποίο στις υποκλοπές είναι απαραίτητο να υπάρχει, είναι νόμιμο και βασίζεται θα έλεγα σε ε, διαφανή θεμέλια νόμιμης πρακτικής υπάρχουν συγκεκριμένοι ε, μέθοδοι. Καταρχής θα πρέπει να, καταρχάς θα πρέπει να εντοπιστεί ένα συγκεκριμένο ε, υποκείμενο το οποίο θα πρέπει ε, να παρακολουθηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Εμείς δεν ψάχνουμε δεξιά-αριστερά ψάχνοντας για συγκεκριμένες λέξεις οι οποίες παρουσιάζουν κινδύνους ή για κάποια ονόματα. Ξεκινάμε ψάχνοντας όμως το τηλέφωνο συγκεκριμένων προσώπων, σύμφωνα πάντα με τις νομικές ρυθμίσεις οι οποίες ισχύουν στις συγκεκριμένες χώρες στις οποίες γίνεται η υποκλοπή. Εμείς δεν συνεργαζόμαστε συστηματικά με τις ε, υπηρεσίες επιβολής του νόμου και δεν έχουμε συστήματα υποκλοπών πέρα από αυτά τα οποία επιτρέπουν οι νομικές ρυθμίσεις κάθε χώρας. Μετά από τη δημιουργία μας σαν επιχείρηση το 2007 φύγαμε από το σύστημα παρακολούθησης και τον Μάρτιο του 2009 σταματήσαμε να ασχολούμεθα με τέτοια θέματα ε, πριν από τις εκλογές στο Ιράν. Το σύστημα παρακολούθησης που είχε ε, δοθεί στο Ιράν το 2008 είναι κάτι το οποίο δεν συντηρούμε, δεν θα συνεχίσουμε εμείς ε, να ασχολούμεθα με τα θέματα αυτά παρά μόνο στα δίκτυα τα οποία εμείς οικοδομούμε. Σχετικά τώρα με τη λειτουργία αυτών των κέντρων στο Ιράν, έπρεπε είναι αλήθεια να καταλάβουμε τα προβλήματα στο Ιράν καλύτερα και περισσότερο θα έλεγα προληπτικά. Υπήρξαν αξιοπιστίες από το Ιράν ότι χρησιμοποιούνται οι τηλεπικοινωνίες σαν μέσο καταστολής της διαφορετικής άποψης και της ελευθερίας λόγου. Λυπούμεθα για τη χρήση αυτή της τεχνολογίας, η οποία τεχνολογία πρέπει μόνο να ωφελεί τον κόσμο ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν λειτουργήσε. Δεν μπορούμε τώρα να επανεφεύρουμε την ιστορία και να την ξαναγράψουμε, αλλά μπορούμε να αποφύγουμε τα λάθη αυτά στο μέλλον. Αξιολογούμε τις πολιτικές μας και τις πρακτικές μας, συνεργαζόμαστε με σημαντικούς εμπλεκομένους, ε, στην περίπτωση αυτή όπως εσείς εδώ σήμερα. Ο στόχος μας είναι οι πολιτικές μας να επανεξεταστούν και να επανεγκριθούν μέχρι τέλος Ιουλίου από το κέντρο ελέγχου της επιχείρησής μας. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να βιαστούμε για να σεβαστούμε μια προθεσμία. Πρέπει να είμαστε σίγουροι. Είναι πρόωρο θα έλεγα οι πολιτικές αυτές να ανακοινωθούν σήμερα αλλά βασίζονται σε συγκεκριμένες αξίες. στις αξίες της διακήρυξης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της ελευθερίας λόγου, της ελευθερίας επικοινωνίας και αυτό χαρακτηρίζει την επιχείρησή μας. Τα δίκτυα τηλεπικοινωνίας ε, στηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της ελεύθερης έκφρασης, της ανταλλαγής απόψεων και της οικονομικής ανάπτυξης. Εμείς ε, έχουμε ευθύνες σαν Nokia Siemens να βοηθήσουμε έτσι ώστε οι τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών τις οποίες παρέχουμε χρησιμοποιούνται για να υποστηρίζουν και όχι να παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η κατάχρηση των τηλεπικοινωνιών είναι κάτι το εντελώς λανθασμένο και όσοι την διαπράττουν θα πρέπει να είναι υπόλογοι για τις δράσεις τους. Ακριβώς στα πλαίσια της τεχνολογικής καινοτομίας και ακριβώς στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξης της τεχνολογίας απαιτείται να υπάρξει μια συνένεση πολιτική σε επίπεδο επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον τομέα αυτό και όχι απλές τεχνικές λύσεις. Είναι σαφές ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και στα οποία αναφερθήκατε δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να επιληθούν. Το ότι τα συστήματα τα οποία παρέχουμε στο Ιράν έπρεπε να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τον τρόπο ο οποίος προβλέπεται από τις διεθνείς νομικές ρυθμίσεις. Συνεπώς λοιπόν εμείς τις ρυθμίσεις αυτές κατηγορούμε ότι δεν τις σεβαστήκαμε. Όπως σας είπα το θέμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις τις οποίες, που παρουσιάζουν δυσκολίες. Ας πούμε υπάρχει το τι είναι το φίλτρο περιεχομένου, το κατάλληλο και ακατάλληλο, στη συγκεκριμένη περίπτωση φίλτρο περιεχομένου. Ας πούμε υπάρχουν κάποια μέσα, κάποια φίλτρα που χρησιμοποιούνται για να απομακρύνονται κάποιοι κίνδυνοι όπως το λεγόμενο spam ή και οι διάφοροι ΙΙ. E e. Αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρείται θεμητό. Υπάρχουν άλλα φίλτρα τα οποία δεν θεωρούνται θεμητά. Πολλές φορές έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις περιπτώσεις των τοπικών νομικών ρυθμίσεων οι οποίες επανειλημμένα είναι ασύμβατες με τις γενικότερες ε, διεθνώς ισχύουσες ρυθμίσεις. Εμείς προσπαθούμε να εντομίζουμε καταστάσεις ε, οι οποίες ε, θα δημιουργήσουν προβλήματα στην χρήση των τεχνολογιών τις οποίες παρέχουμε έτσι θα μπορέσουμε να επιλέξουμε το ποιες είναι οι τεχνολογίες οι οποίες είναι οι κατάλληλες για κάθε χώρα και θα πρέπει να αναζητήσουμε και μεθόδους για να μετριάσουμε τους κινδύνους και τις συνέπειες που μπορεί να προκληθούν και όχι να εμείνουμε σε συγκεκριμένες προθέσεις μάλλον, δηλώσεις προθέσεων, χωρίς να πάρουμε κάποια απτά μέτρα το περιβάλλον ανθρώπινα δικαιώματα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα που ισχύει σε μια χώρα μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό το βιώσαμε κατά τη διάρκεια της διάρκειας ζωής των συστημάτων μας. Εμείς αναπτύξαμε ας πούμε δίκτυα σε μια κυβέρνηση η οποία ήταν φυσιολογικό να το κάνουμε κάποτε και σε κάποια άλλη φάση κάτι τέτοιο αυτό ήταν πλέον απαράδεκτο. Δεν θα ήθελα να κάνω συστάσεις σε λήψη χρόνου. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που λέτε ότι μάθατε από την εμπειρία σας και ξανασκέφτεστε τα πράγματα μαζί με τους, ε, με τους διάφορους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και ημών εδώ. Για να δούμε τώρα η Google τι κάνει. Ο κύριος Σάιμον Χάμπτον είναι εδώ Διευθυντής για τη Δημόσια Διοίκηση. Ευχαριστώ. Μεγάλη χαρά που είμαι εδώ σήμερα. Μου ζητήθηκε να μιλήσω λίγο για την Κίνα. Και να πω και κάποια πράγματα για την πολιτική της Google. Σκέφτηκα να ξεκινήσω με την Κίνα για το τι έγινε στην αρχή του χρόνου. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα ανακαλύψαμε ότι υπήρχε μια ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου επίθεση στο, στην υπηρεσία του Gmail μας. Εμείς και άλλες 20 εταιρείε ε, από την ε, απίθεση αυτή και επίσης ανακαλύψαμε ότι οι χρήστες του Gmail επίσης ε, είχαν υποστεί τέτοιες ε, επιθέσεις ε, phishing που ήταν ας διάφοροι που προσπαθούσαν να εκμεύσουν πληροφορίες από αυτούς. Είδαμε λοιπόν ότι υπήρχε μια τάση να, όλοι αυτοί να εμπλέκονται συχνά σε διάφορες ε, εκστρατείες για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα. Από τους Ολυμπιακούς Είδαμε ότι αυξήθηκε η λογοκρισία και η πίεση. Μας κατηγόρησαν ότι είμαστε στην, επίχει, στην βιομηχανία της πορνογραφίας. Αυτή ήταν και η δικαιολογία που χρησιμοποιήθηκε για να ε, περιορίσουν ε, τα προϊόντα στην, ε, στις μηχανές αναζήτησης. Το Μάρτι Από τους ρεπόρτους χωρίς σύνορα είπαμε ότι η υπηρεσία CN που, ήταν στην, ε, που δραστηριοποιείται στην ε, Κίνα ε, μπόρεσε να διεξάγει τις υπηρεσίες της χωρίς λογοκρισία. Οι χρήστες μας συνεχίζουν να βλέπουν ότι κάποιες μέρες έχουν πρόσβαση, κάποιες δεν έχουν στις υπηρεσίες που δεν την χάνουν λογοκρισίας. Κάποιες φορές αυτό που ψάχνουν ε, δεν μπορούν να το βρουν. Μπορέσουμε κάποιος να ψάξει να αναζητήσει κάτι πολύ ας πούμε συνηθισμένο και να βρει κάτι ως αποτέλεσμα, αλλά κάτι που να είναι πιο ευαίσθητο δεν του το βγάζει. Γιατί το firewall είναι πάρα πολύ ευαίσθητο για τα θέματα αυτά. Το YouTube ας πούμε δεν είναι διαθέσιμο στην Κίνα προς το παρόν και για αρκετούς μήνες δεν είναι διαθέσιμο. Αυτό που κάνουμε είναι να είμαστε πολύ διαφανείς, οπότε μπορεί κανείς να πάει στη Google, στη σελίδα μας, google.com κάθετος PRC, κάθετος report και να δει ποιες είναι οι ε, υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες και ποιες δεν είναι στην Κίνα. Για τις ε, επιχειρήσεις μας, από την λήψη της απόφασης, είδαμε ότι ε, η βασική μηχανή αναζήτησης, αναζήτησης έχει αυξηθεί ε, εμείς έχουμε χάσει 5% περίπου της, ε, του πεμεριδίου αγορά στην Κίνα και η Μπάιντο και κάποιοι άλλοι ανταγωνιστές από τη ΣΥΠΑ έχουν καταφέρει να πάρουν με, το μέρος τους κάποιους από τους ε, δικούς μας μηχανικούς ώστε να, πάνε στην, να δουλέψουν για αυτούς. Τώρα, πώς απαντούμε εμείς. Καταρχήν, για την ασφαλεία και την ιδιωτική σφαίρα αναζητήσεις χρησιμοποιώντα το κρυπτογραφημένο, τη κρυπτογραφημένη δυνατότητα με το HTTPS. Μπορεί κανείς τώρα να ψάχνει μέσω αυτού του συστήματος. Οπότε είναι σχεδόν αδύνατο να ψάξει κανείς και να βρει τι αναζητάει ο κάθε Βεβαίω, εντάξει, μπορεί να μπλοκάρει την πρόσβαση στο HTTPS, αλλά εν πάση περιπτώσει εμεί έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα που να μπορεί να αναζητεί κανεί ό,τι θέλει μέσω του HTTPS. Επίση, πρέπει να δούμε τον όλο τομέα τη ασφάλεια στι ε, υπηρεσίε στο ίντερνετ. Και επίσης κοινοποιήσει για παραβάσεις είναι πολύ σημαντικέ. Δεχτήκαμε ότι ε, εντάξει, ε, συνέβησαν αυτές οι επιθέσεις. Άλλες 20 εταιρείε υπέστησαν τέτοιες επιθέσεις, ε, αλλά δυστυχώς δεν τις έχουν ανακοινώσει αυτές τις πληροφορίες, ενώ εμείς το κάναμε. Επίσης, πρέπει να δούμε λίγο τα του οίκου μας. Εντάξει, καλό, ένα πράγμα είναι να κριτικάρουμε τους Κινέζους, αλλά ένα πράγμα είναι να δούμε τι κάνουμε και γενικώ στον υπόλοιπο κόσμο. Ε, γι' αυτό έχουμε εισαγάγει αυτή την πτυχή της διαφάνειας, για να απαντήσουμε και στα αιτήματα που λάβαμε από διάφορες κυβερνήσεις ανά τον κόσμο Πάλι μπορείτε να πάτε στην ε, σελίδα μας ε, google.com κάθετος government requests και να δείτε ποιες είναι οι αιτήσει που έχουμε λάβει από διάφορες χώρες του κόσμου, από διάφορες κυβερνήσεις για να ε, μειώσουμε την πρόσβαση σε συγκεκριμένα περιεχόμενα. Ξεκινήσαμε λοιπόν μια τέτοια συζήτηση για όλο αυτό τον τομέα της Παρέμβαση των κυβερνήσεων ε, που ζητούν από τέτοιες υπηρεσίες, ε, εταιρείες τεχνολογίας να λάβουν τέτοια δράση. Αυτό το θέμα βέβαια δεν θα ολοκληρωθεί άμεσα, γιατί βασίζεται σε δύο οικονομικές τάσεις. Καταρχήν η παγκοσμιοποίηση και η ε, μετάβαση στην, στην οικονομία της γνώσης. Οπότε πάντα θα βρισκόμαστε στην Ευρώπη ε, λειτουργώντας μέσα σε έναν, με έναν οικονομικό τρόπο, προσπαθώντας να επιτύχουμε την, ε, να επενδύσουμε στη γνώση. Και από τον τομέα των υποδομών και για τον τομέα των υποδομών είναι σημαντικό αυτό. Οπότε ένας από τους τρόπους που προσπαθήσαμε να λύσουμε το θέμα, όπως είπε και ο Άντριο πιο πριν, είναι η πρωτοβουλία για τα Global Networks. Μια πρωτοβουλία τριών εταιριών, online, δεν είναι μίας οργάνωσης. Η Google, η Microsoft και η Yahoo με, μαζί με διάφορες μη κυβερνητικέ οργανώσεις δημιούργησαν έναν κώδικα δοντολογίας και εδώ στον τομέα αυτό θα θέλαμε να ε, μπλακούν ε, και οι Ευρωπαίοι φορείς. Είναι σαφές ότι ο κώδικας θα πρέπει να αναθεωρηθεί, να αντικατοπτρίζει όλα όσα αφορούν τις υπόλοιπες εταιρείε ε, που δεν λειτουργούν με τον ίδιο ακριβώ ε, στόχο όπως οι τρεις που έφτιαξαν τον κώδικα. Αλλά γενικώ ε, η αυτορύθμιση είναι συνήθως καλή για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα στο ίντερνετ. Και επίσης υπάρχει συγκεκριμένο πεδίο για τη συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και ΕΥΠΑ ΕΕ στον τομέα αυτό. Μας υποστήριξαν πάρα πολύ διάφοροι, διάφοροι εταίροι, ε, επιχειρήσεις. Η συζήτηση λοιπόν αυτή δεν νομίζω ότι θα κλείσει σύντομα και ελπίζω να μπορέσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο να πιέσει περισσότερο στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας εξηγήσατε κύριε Χάμπτον και τώρα ε, μπορούμε να τα ξαναδούμε όταν αρχίσει η συζήτηση και το κύριο Σούσο. Δεν ελπίζω δεν κρυούργη κατά κάποιο από το όνομά σας, είναι ο υποδιευθυντής της ε, Global Freedom Consortium και θα μας μιλήσει για τη νέα, τις νέες μορφές της ε, τηλεόρασης και θα μας μιλήσει και με τη λογοκρισία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ την Επιτροπή σας και εσάς που μας καλήσατε για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα της ε, πληροφορικής και των δικαιωμάτων. Να δούμε συγκεκριμένα τι ισχύει στην Κίνα. Η Κίνα είναι παράδειγμα προς αποφυγή όσον αφορά το συστηματικό λόγο του διαδικτύου δεκάδες των χιλιάδων ε, αστυνομικών ασχολούνται με αυτό. Ο κόσμος πάει στη φυλακή γιατί εκφράζεται μέσω του ίντερνετ. ΣΥΣΚΟ και άλλες ε, εταιρείε φιλτράρουν ό,τι η κυβέρνηση θέλει. Και αυτή η διαδικτυακή λογοκρισία έχει πάει και σε άλλες χώρες τώρα, έχει μεταδοθεί Μπούρμα, Κούβα, Ιράν και στην Κεντρική Ασία, πρώην Σοβιετικής Δημοκρατίας, όλα ένα και περισσότερο μιμούνται τέτοιες ε, μεθόδους για να ελέγξουν την πληροφόρηση και να μην αφήσουν τον κόσμο να επικοινωνεί με τις υπόλοιπες προς την υπόλοιπο κόσμο. Αυτό είναι το φαινόμενο του 21ου αιώνα και αυτή, αυτός ο έλεγχος της ε, πληροφόρησης γίνεται για λόγους προπαγάνδας, όποτε έχουμε κάποια κρίση στην ε, χώρα. Ε, όλα τα ΜΜΕ τα ρίχνουν στην ε, Δύση να δικαιολογήσουν την κυβέρνηση. Το 2008 το ίδιο έγινε και με τα γεγονότα στο Θιβέτ. Είχαμε και και για όλα, και όλα κατηγορήθηκαν οι δυτικέ εταιρείε όπως η Καρφούρ. Το ίδιο ισχύει και για ε, διάφορα σκάνδαλα, διάφορες ε, επιδημίες και όλα είναι και περισσότερο επομένως κατηγορείται η Δύση. Κλειστή κοινωνία, λογοκρισία Όμως υπάρχει κάποια ελπίδα, υπάρχουν κάποια συστήματα κατά της ε, λογοκρισίας όπως αυτό το βήκαν το δικό μας κονσόρτσιουμ οπότε κατά αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουν την στο ίντερνετ. Ε, Αμερικάνοι μηχανικοί έχουμε δουλέψει για αυτά τα μέτρα λογοκρισίας και ο, ομιλητής επίσης. Κάποιοι από εμά ήμασταν ε, στην σφαγή της Τιανανμένη ε, το 89. Είδαμε πως ε, στρέβωσαν την αλήθεια οι αρχές. Το 99 επίσης, με την επίθεση κατά των Φαλαγκόγκ, ε, είχαμε και εκεί φαινόμενα προσπάθειας στρέβλωσης της κοινής γνώμης. Ακολούθησαν συλλήψεις, δίκες, διώξεις ένας φίλος μου φωνεύτηκε όσο ήταν ε, ε, κρατούμενος σε φυλακή της Σαϊγκόν και εξάδελφος σε καταναγκαστικά έργα στην Κίνα. Πιστεύουμε ότι η ελεύθερη ώρα της πληροφορίας είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να ανοίξει μια κλειστή κοινωνία και να προστατευτούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι πολιτικές ελευθερίες. Γι' αυτό και ξαγρυπνήσαμε πολλές φορές, πολλά βράδια, ώστε να μπορέσουμε να παρακάμψουμε τους λογοκριτές, τους Κινέζους και άλλους. Και έτσι να είναι δυνατή η επικοινωνία από και προς την Κίνα. Όλοι στην EJIF ουσιαστικά από το στέρημά μας προωθούμε τους σκοπούς της εταιρεία, αλλά δεν χρεώνουμε τους χρήστες των συστημάτων μας. και προσπαθούμε να αλλάξουμε τις ε, διευθύνσεις των σερβερ που έχουμε για να μην υποστούμε την ε, λογοκρισία. Κάθε κλειστή κοινωνία στον κόσμο έχει προσβασιμότητα στους δικούς μας σερβερς. Κίνα και Ιράν, αλλά και Μπούρμα εξοχήν είναι χώρες όπου υπάρχει κόσμος τέτοιος. Μέσα του σέρβου μας περνάει όλη τους η επικοινωνία. Τέλος Αυγούστου 2007 στην Μπούρμα επίσης είχαμε φαινόμενα καταστολής και πάρα πολλοί Μπουρμέζοι ε, μετέδωσαν τα γεγονότα μέσω των δικών μας συστημάτων. και φυσικά η κυβέρνηση της χώρας έκανε προσπάθειες να φημώσει αυτούς τους ε, αντιπολιτευόμενους. Οπότε έχουμε κάποια κρίση που παρουσιάζονται οι ροή πληροφοριών προσφέρει και 400 φορές. Ε, όπως έγινε και στο Ιράν πέρσι τον Ιούνιο είχαμε εκεί 600% αύξηση του, της, ε, της λειτουργίας του, της επικοινωνίας μάλλον μέσα σε μια εβδομάδα. Ένα εκατομμύριο ήταν οι Ιρανοί που χρησιμοποίησαν τα συστήματά μας για να επισκεφθούν το Facebook και άλλα συστήματα. Twitter, Google, YouTube. Και ε, έτσι δημοσίευσαν ε, πληροφορίες, ε, φωτογραφίες για τα μέτρα καταστολής. Όταν επομένως δοκιμάσουν την ελευθερία αυτή που είναι μια κλειστή κοινωνία, τότε θα σταματήσουν να σκύβουν το κεφάλι. Ακριβώς αυτό έγινε και στην Ανατολική Ευρώπη. Και η μάχη ήταν για την πληροφορία και τώρα είναι για, τις, ε, για, για πόρους. Γιατί προσπαθούν να μας μπλοκάρουν με κάθε τρόπο. Άρα θα πρέπει η προτεραιότητα είναι να εξασφαλίσουμε την ελευθερία της επικοινωνίας με το ίντερνετ για αυτές τις κλειστές κοινωνίες. Παντού στον κόσμο. Και θα πρέπει σε προσπάθειες που γίνονται για την υπεράσπιση του Ιντερνετ και αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να υπάρχει προστασία και ενίσχυση. Όπως σε Κίνα και σε Ιράν λοιπόν έχουμε καταστολή και το πρόβλημα της ε, λογοκρισίας δεν είναι μόνο εσωτερικό σε αυτές τις χώρες μόνο γιατί από πρώτο χέρι έμαθα τι θα πει κινέζικη λογοκρασία όταν ε, ένα κινέζικο ε, κανάλι δορυφορικό φημώθηκε από τους Κινέζους. Ε, έκλεισαν τον γαλλικό δορυφόρο. Είχαμε μόνο μια τηλεόραση που χωρίς λογοκρισία μετέδιδε και ποτέ δόθηκε ικανοποίηση γιατί κόπηκε το σήμα αλλά από ό,τι φάνηκε ήταν πολιτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διαχείρισης του Δορυφόρου για να ικανοποιήσει και να ευχαριστήσει τους Κινέζους. Η Eurosat συγκεκριμένα. Το ίδιο έγινε και στον Κάφκασο. Η γεωργιανή τηλεόραση εξέπεμψε στα ρωσικά. Η Γκασπρόμ και, και, οι Ρώσοι γενικότερα θέλανε αυτό να το φρενάρουν, αλλά ευτυχώς υπήρξε προστασία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υπήρξε πίεση να αφαιθεί ελεύθερη αυτή η εκπομπή και όπως ε, είχαμε μετά την συνήθεια της Αβώνας και κατοχυρώθηκε η ελευθερία της έκφρασης και της πληροφορίας ελπίζουμε ότι έτσι τώρα το κοινοβούλιο θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ελευθερία για τα μέσα ενημέρωσης Κομισιόν και Συμβούλιο θα ακολουθήσουν. Η τηλεόρασή μας ήταν μια χτίδα ελπίδας. Όπως ακριβώς ήταν και για την Ανατολική Ευρώπη η Αμερικανική τηλεόραση. Χρησιμοποίησαν το φαξ στη Σοβιετική Ένωση ε, για, για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν, για να μπορέσουν να πούν τι, τι συνέβαινε εκεί. Και, και τελικά γκρεμίστηκε το παραπέτασμα. Τώρα έχουμε το Ιντερνετ, έχουμε και άλλα μέσα για ελευθερία έκφραση. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ελπίδα για ελευθερία και δημοκρατισμό και για την ε, εξέλιξη της κοινωνίας. Θα ήταν ε, έτσι καλύτερο καλύτερος κόσμος αν όλοι μπορούσαμε να συνοηθούμε, αν δεν είχαμε πια καταστολή, ολοκληρωτισμό και Πρετάνευε η ελευθερία σε όλες τις κοινωνίες. Σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Η Αντιπρόεδρος, κυρία Αντρικένε, και άλλοι συνάδελφοι, ε, καταλάβαμε τι είπατε όταν μας είπατε για τη Γιούτελσατ, γιατί με τους δημοσιογράφους χωρίς σύνορα και με άλλους είχαμε ε, αναλάβει τη σχετική πρωτοβουλία τότε. Σήμερα, πάντως, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία υπαρχής σε σχέση με το πώς έγινε και κόπηκε το σήμα το δορυφορικό μεταξύ Utelsat και αυτών των ε, εταιριών τηλεοράσεων. Παραμένει λοιπόν το ερωτηματικό και θυμάμαι και το κανάλι του Κάφκασου, τώρα το εμποροδικείο στο Παρίσι, διερευνά τι έγινε, αν υπάρχουν κάποια παραβιάσεις του δικαίου, εμπορικού δικαίου, τέλο πάντων. Διερευνάται το θέμα, εκκρεμεί ενώπιον του δικαστήριου και ευχαριστούμε για το σημασία μα είπατε όσον αφορά την ελεύθερη τη πληροφορία για κάποιε χώρε όπω το η Κίνα και το Ιράν. Ακόμη, δύο έχουν ζητήσει το λόγο. Και έχουμε μισή ώρα για, για απαντήσεις. Και τώρα το ρόλο έχει ο κύριος Μακιγιάμα. Ο κύριος Μακιγιάμα είναι επισκέπτης καθηγητής Ε, ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος στην Σουηδία και μπορείτε να μας μιλήσετε για περίπου 5 λεπτά όσον αφορά την εμπορική πολιτική, την λογοκρισία και δίνουμε τη σκητάλη στον κύριο Μάκη Γιάννα. Madam Chair, member of the subcommittee, thank you. Πρόεδρε, ευχαριστώ που οργανώσατε αυτή την ακρόαση. Χασόκλη Μακιγιάμα ονομάζομαι. Economy. Uh, I have been asked today to testify on internet Ασχολούμαι με τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ίντερνετ. Μιλάει πολύ γρήγορα ο κύριος. Και του γίνεται μια σύσταση να μιλάει λίγο πιο αργά. Η λογοκρισία στο διαδίκτυο είναι όντως περίπλοκο θέμα και στην Κίνα είναι το πιο περίπλοκο θέμα που υπάρχει. Πιο περίπλοκο από ό,τι πουθενά αλλού. Γιατί το ίντερνετ είναι τελείω διαφορετικό στην Κίνα από ό,τι σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Πάνω από 18.000 ιστοσελίδε, οι περισσότερες είναι συνηθισμένε και είναι μπλοκαρισμένε όλες στην Κίνα. Και όταν είναι κανεί εκεί, και οι τοπικές ιστοσελίδε και οι ε, αλλοδαπές ε, πρέπει να επιδεικνύουν κάποια πειθαρχία που είναι έτσι κατεφημισμόν η λογοκρισία. Επίσης πρέπει να πω ότι υπάρχουν ε, μεγάλες διακρίσεις, ε, ε, μπλοκάρονται στο σελίδες χωρίς κανέναν λόγο, ε, υπάρχει μεγάλη καθαριστέρηση στο να φορτώσει μια σελίδα ώστε να είναι τελείως άχρηστη, ε, καταραίουν οι σερβερς, Η Κίνα σήμερα είναι η μεγαλύτερη online αγορά. 338 εκατομμύρια χρήστες του ίντερνετ, ενεργοί χρήστες. Έχει ξεπεράσει τις ΗΠΑ και είναι η δεύτερη, παγκόσμια, δεύτερη μεγαλύτερη παγκόσμια οικονομία. 70 εκατομμύρια blogs υπάρχουν στην Κίνα. Πολλά ε, δίνουν πολύ πλουραλιστικέ ιδέες για τους, ε, τοπικές, για τους τοπικούς άρχοντες, για τις εταιρείε ε, και για διάφορους, διάφορες κάποιες νομοθεσίες που, είναι, που δεν είναι πολύ φιλικές προς, το, προς τους πολίτες. Η... Τα κινέζικα προϊόντα έχουν καταλάβει τον κόσμο. Έχουμε ακούσει και από την, από την Google διάφορα παράπονα για το τι γίνεται στην ε, Κίνα. Η Baidu είναι μια μεγάλη ας πούμε μηχανή αναζήτησης ε, η οποία έχει ξεκινήσει δραστηριότητα και στο εξωτερικό. Ο οικονομικός προστατευτισμός επίσης είναι σημαντικό θέμα για την ε, λογοκρισία που υπάρχει στην Κίνα. Η νέα βιομηχανική πολιτική για την Κίνα θέλει να αποδεσμεύσει τον, ε, την Κίνα από την, την υπόλοιπη παγκόσμια οικονομία. Η Κίνα προσπαθεί να εφαρμόσει περιορισμούς σε προϊόντων πληροφορικής ε, που, τα οποία ε, παράγουν μόνο η ντόπιοι παραγωγοί. Εγώ θεωρώ ότι τα θέματα ανθρωπινών δικαιωμάτων θα πρέπει να υποστηριχθούν. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι το να θέσουμε μέσω, τα, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω εμπορικής πολιτικής είναι αντιπαραγωγικό και αναποτελεσματικό. Αλλά το θέμα της λογοκρισίας στην Κίνα είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό γιατί η κινητοποίηση και η πραγματική φύση της ε, λογοκρισίας είναι εμπορική. Ενώ υπάρχουν διάφοροι φορείς που ακούσαμε σήμερα, και υπάρχουν και τα φόρουμ στον ΟΗΕ, οι διάφοροι φορείς του ΟΗΕ, όπως το Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Συμβούλιο Διακυβέρνηση, δίνουν το σωστό πολιτικό περιθώριο για να αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό. Υπάρχουν όμως και άλλοι φορείς, ο ΠΟΕ α πούμε, όπου η Κίνα προσχώρησε το 2001, Εκεί μπορεί η Κίνα να λύσει τα προβλήματά της τα εμπορικά με τα κράτη-μέλη και η προσχώρηση στον ΠΟΕ έχει δεσμεύσει την Κίνα σε απεριόριστη πρόσβαση ε, στην αγορά των, ε, των ε, υπηρεσιών online στις υπόλοιπες χώρες. Στις αγορές δηλαδή των υπόλοιπων χωρών. Η Κίνα παραβιάζει αυτή την πρόσβαση για προϊόντα πολιτισμού όπως η μουσική εδώ το πάνελ λέει ότι η λογοκρισία στην Κίνα ήταν δυσανάλογη σε σχέση και με το ηθικό επίπεδο που, ήθελαν να θέσουν, που ήθελαν να θέσουν στην Κίνα. Οπότε υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήματα για να λυθεί το θέμα αυτό της λογοκρισίας και σε σχέση με τον ΠΟΕ, διότι θα έχει καταρχήν αποτελέσματα. Η Κίνα έχει δείξει ότι θα συμφωνήσει, θα συμμορφωθεί με τους κανόνες, με τους οποίους βεβαίως ε, διαφωνεί κάθετα. Δεύτερον, ο ΠΟΕ είναι μη πολιτικό φόρουμ. Η Κίνα καταλαβαίνει ε, πώς ε, λειτουργούν οι διαπραγματεύσεις, σέβεται τον ΠΟΕ και επίσης ε, χρησιμοποιεί τους κανόνες ε, η Κίνα έχει φέρει δύο, δύο υποθέσεις ενώπιον της, του ΠΟΕ εναντίον της Ευρώπης και η Ευρώπη τέσσερις εναντίον της Κίνας. Επίσης η Κίνα υπάρχει, έχει μπει σε πολλές ε, διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα, μπορέσει να, θα μπορέσουν έτσι να τεθούν κάποιοι διεθνείς κανόνες ε, και από τις επιχειρήσεις και από τις μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις για τα καταχρηστικά οικονομικά μέτρα, ώστε να ενισχυθεί ο ΠΟΕ και η πολυμερής, το πολυμερές σύστημα στο οποίο έχει εμπλακεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μειωθεί, θα απαλληφθεί η λογοκρισία. Η υπόθεση όμως του ΠΟΕ έχει και κάποια όρια. Αντιμετωπίζει μόνο το δικαίωμα των ξένων στο σελίδο να μπουν στην Κίνα και προστατεύει, ε, τους προστατεύει από το μπλοκάρισμα, αλλά δεν προστατεύει τις, ε, τις επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών στην Κίνα, τις τοπικές. Επίσης, ε, χώρες όπως η Ρωσία, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα δεν είναι μέλη του ΠΟΕ, οπότε δεν επηρεάζονται από τους κανόνες. Στην περίπτωση όμως της Ρωσίας και του Ιράν, οι συνεχιζόμενες ε, ε, διαπραγματεύσει για την προσχώρηση δεν μπορούσαν να είναι η ευκαιρία για να γίνει η μεταρρύθμιση. Παρά λοιπόν τα προβλήματα, ο ΠΟΕ όντω ε, είναι, αρκετά, είναι το σωστό φόρουμ σε αντίθεση με άλλα. Και θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερο από τα μονομερή μέτρα που έχουν ληφθεί κατά καιρού. Οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα, θα περιόριζαν τις, ε, το εμπόριο των επιχειρήσεων με την Κίνα ή με άλλες βολιταρχικές χώρες ή θα ποινικοποιούσαν τις, ε, και η Κίνα θα ποινικοποιούσε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εναντίον των δικών της. Οι υπηρεσίες online και οι τηλεπικοινωνίες ε, είναι τεχνολογίες που απελευθερώνουν που, δεν θα, που θα μπορούσαν να ε, βοηθήσουν στην ε, μείωση των ε, ιστοσελίδων που μπλοκάρει η Κίνα. Το ερώτημα λοιπόν είναι πού βάζουμε το όριο. Η τεχνολογία του ίντερνετ μιλά για καθημερινά προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς και λόγους. Αν μπορώ τώρα να κάνω εγώ έτσι μια ανάλυση, ίσως να, είναι, να μιλούμε για μια υπόθεση όπου θα μπορούσε κανείς ε, να κατηγορήσει την, ε, την Κίνα για, για πολλά πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλές αποδείξεις και θα ήθελα εγώ να ενθαρρύνω και τα κρατημέλη και την Κομισιόν να κάνουν τα απαραίτητα βήματα, να ζητήσουν διαβουλεύσεις, ίσως να κάνουν και μια ε, παρέμβαση στον ΠΟΕ για το θέμα της Κίνας. Ευχαριστώ. This Πράγματι προκλητική η παρουσίασή σας. Έχουμε τον κύριο Τίμανς από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα, τον οποίο έχουμε τακτικά θα έλεγα εδώ. Ακούσαμε πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες. Θα ήθελα να μπορέσετε να σχολιάσετε για το τι θα μπορεί να κάνει στα πλαίσια και του πλαισίου του ΠΟΕ η Ευρωπαϊκή Ένωση, Μια και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνη για την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα εμπορικά φόρα. Δεν νομίζω ότι θα περιμένετε να έχουμε ήδη χωνέψει σε εισαγωγικά όλες αυτές τις καινοτόμες απόψεις και τολμηρές απόψεις που ακούστηκαν κυρίως από τον καθηγητή κύριο Πούντενφατ. However, that I uh, was also quite attentively listening to all the statements which have been made. I apologize for having... Συγγνώμη που ήρθαμε Ήρθα καθυστέρηση, αλλά συμμετείχα σε διεθνείς διαπραγματεύσεις και δεν μπορούσα να φύγω νωρίτερα. Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν τεράστια προβλήματα, τεράστιες προκλήσεις καλύτερα και τεράστιες ευκαιρίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο χρήστης του ίντερνετ και ο λογοκριτής σε πολλές χώρες είναι σε μία μόνιμη μάχη του ποιος θα αποδειχθεί πιο έξυπνος χρησιμοποιώντας ε, το σωστό λογισμικό και το σωστό υλικό επίσης έτσι ώστε να μπορέσουν οι χρήστες να αποφύγουν κάποια από τα μέσα καταστολής. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο, πολύ πιο δύσκολο πια ε, για τα ολοκληρωτικά καθεστώτα να καταστήλουν την ελεύθερη έκφραση μέσω της πλήρους κατάργησης της πρόσβασης ε, στο διαδίκτυο. Ακόμα και στην Κίνα, παρά αυτά τα οποία ακούσαμε προηγουμένως, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ταυτόχρονα όμως οι σύγχρονες τεχνολογίες ενισχύουν ε, τις ελεγκτικές ικανότητες των κυβερνήσεων. Η έκθεση επιστεί την προσοχή μας στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα μέσα της τεχνολογίας για να καταστήλουν την επικοινωνία και μέσω ε, των τηλεπικοινωνιών του Twitter κτλ. Όλοι ενθυμούμεθα επίσης τα πάρα πολύ μικρά βίντεο τα οποία είδαμε τον προηγούμενο Ιούνιο από την Τεχεράνη τα οποία είχαν ε, ληφθεί από τα μικρά κινητά τηλέφωνα και τα οποία μετέφεραν αυτή την ακνόσφαιρα τρόμου. Οι μηχανισμοί ελέγχου λοιπόν είναι όλο ένα και πιο αόρατοι, παρακολουθούν τις επικοινωνίες και να ανοιχνεύσουν τις ε, επικίνδυνες ενέργειες. Η έκθεση αναφέρεται και σε άλλα δύσκολα προβλήματα όπως το πώς να εξισορροπήσει κανείς τα δικαιώματα των προσώπων, την πρόσβασή τους στη γνώση και τη συμμετοχή τους στην πολιτιστική ζωή σε σχέση με την προστασία των, ε, της πνευματικής ιδιοκτησίας ή επίσης την ανάγκη καταπολέμησης του αποκλεισμού των φτωχών μειονοτήτων και την πλήρη πρόσβασή τους στις, στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Γίνονται ορισμένες περίπλοκες συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της έκθεσης που αφορούν πολλούς τομείς της πολιτικής μας. Η σημαντική αυτή έκθεση την οποία συζητάμε σήμερα και η έκθεση στην οποία αναφέρθηκε ο Ευρωβουλευτής Βάγνερ, την οποία δεν γνωρίζω ακόμα, είναι ένα τμήμα θα έλεγα μιας μορφής διαλόγου ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Να προσπαθήσω να αντιδράσω για κάποιες από αυτές τις συστάσεις, αλλά σε εντελώς πρώιμο στάδιο. Αναφέρθηκε στην έκθεση αλλά και ακούστηκε εδώ προφορικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να θέσει το θέμα των ελευθεριών στο ίντερνετ στις διμερείς επαφές που έχουμε στο διμερή διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το κάνουμε αυτό. Ήδη το κάνουμε. Συμφωνώ βέβαια ότι ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι το μοναδικό μέρος όπου μπορούν να τεθούν όλα αυτά τα θέματα και απαιτούνται ταυτόχρονα κάποιες πλέον καινοτόμες και διαφορετικές αντιμετωπίσεις επικοινωνίας έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε όλα τα φόρα στα οποία τίθενται τα θέματα της ελευθερίας έκφρασης όπως επίσης και της χρήσης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Βάγνα ότι θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα διεθνή φόρα όπως επίσης και το Φόρουμ για την διακυβέρνηση του διαδικτύου και να εκφέρουμε συγκεκριμένες και ενιαίες απόψεις σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, επανεξετάζοντας τις θέσεις μας στα πλαίσια του, των Ηνωμένων Εθνών και στα πλαίσια της συμμετοχής μας σε ορισμένες συμβάσεις και να δούμε και την ανάγκη για κάποιες νέες ρυθμίσεις σε διεθνές επίπεδο. Είναι σαφές ότι η διασπορά που χαρακτηρίζει γενικά το θέμα του διαδικτύου δημιουργεί δυσκολίες σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση και απαιτούνται φάνταστες λύσεις. Ξέρω ότι η κυρία Μοριγιόν αναφέρθηκε στην ανάγκη νέων νομοθετικών διεθνών ρυθμίσεων όπως επίσης ε, τις, ε, τους ελέγχους των εμπειρογνωμόνων Ζήτησε η κυρία Μοριγιόν επίσης να συμπεριλαμβάνουν οι εμπορικές συμφωνίες ειδικέ ρυθμίσεις για το διαδίκτυο και για το εμπόριο μέσω διαδικτύου και την ανταλλαγή αγαθών γενικότερα. Θα συμφωνήσω επίσης με τον Μακαγιάμα και άλλους ότι γενικότερα Είμαστε διστακτικοί στο να βάζουμε πάρα πολλούς περιορισμούς στο εμπόριο. Το σκεφτόμαστε. Το οποίο εμπόριο θα πρέπει, σύμφωνα με αυτά που πιστεύουμε, να είναι όσο πιο ανοιχτό γίνεται. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνουμε υπόψη τις υποχρεώσεις με τις οποίες θα πρέπει να δράσουμε στα πλαίσια των συμφωνιών του ΠΟΕ. Υπάρχουν άλλοι τρόποι τώρα για να ρυθμίσει κανείς ε, τα θέματα αυτά. Η μονομερής αντίληψη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων δεν είναι η πλέον πρόσφορη. Έχουμε συζητήσει κάποιες περιπτώσεις συγκεκριμένες και σκεφτόμαστε ίσως θα πρέπει να θέσουμε σαν θέμα στα πλαίσια των επίσημων συνομιλιών μας στο εσωτερικό του ΠΟΕ για το θέμα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και της Κίνας αλλά τίποτα δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, απλά θα ήθελα να πω ότι εξετάζουμε όλες αυτές τις συστάσεις και θα τις εξετάσουμε με σοβαρότητα και σε βάθος. Θα ήθελα επίσης να τονίσω αυτά τα οποία μας έχουν ήδη αναφέρει οι εκπρόσωποι των βιομηχανιών και των επιχειρήσεων για κάποιες εθελοντικές συμφωνίες τις οποίες έχουν κάνει μεταξύ τους οι συμφωνίες αυτές είναι χρήσιμες, οι πρωτοβουλίες αυτές είναι πολύ χρήσιμες και μπορεί κανείς πάνω σε αυτές να βασίσει την περαιτέρω δράση του. Και όπως είπε και ο εκπρόσωπος της Google, το να μπορέσει κανείς να χρησιμοποιήσει την γνώση την οποία έχουν ε, κάποιες επιχειρήσεις ευρωπαϊκές γύρω από αυτό τον τομέα τις καθιστά πολύ χρήσιμες. Γιατί οι ίδιες αντιμετωπίζουν πολλές φορές ιδιαίτερες δυσκολίες. Υπάρχει επίσης και το θέμα του τι μπορείτε εσείς να κάνετε για να προωθήσετε την καινοτομία και την ευκολότερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η έκθεση Pundenfat λέει ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα ταμείο καινοτομία για τις νέες τεχνολογίες που θα υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στον ψηφιακό κόσμο. Όπως ξέρετε, οι οικονομικοί πόροι τους οποίους έχουμε στη διάθεσή μας, ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σχετικά λίγοι. Αλλά θα μιλήσω φυσικά με τους συναδέλφους από τον τομέα της έρευνας και τον τομέα της τεχνολογίας, για να δούμε αν υπάρχουν δυνατότητες ε, να προκαλέσουμε κάποιες αντιδράσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Η έκθεση ζητά επίσης να προχωρήσουμε και σε σεμινάρια προς μεμονωμένα πρόσωπα έτσι ώστε να μπορούν να ξεφεύγουν από τις πιέσεις ε, της ε, καταστολής και της κρατικής παρέμβασης. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε το μέσο για τη δημοκρατία, έχουμε ορισμένα προγράμματα τα οποία είναι ιδανικά θα έλεγα προς την κατεύθυνση αυτή και τα οποία θα επιτρέψουν στους εταίρους μας να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα θέματα με καλύτερο τρόπο. Ας κλείσω λέγοντας ότι ακούσαμε μία σειρά από απόψεις οι οποίες πρέπει να εξεταστούν σε βάθος στο εσωτερικό των υπηρεσιών της Επιτροπής. Θα προσπαθήσουμε να διασταυρώσουμε την εμπειρογνωμοσύνη πολλαπλών υπηρεσιών και να δούμε τι συνέχεια μπορούμε να δώσουμε προς την κατεύθυνση αυτή προσωπική μου άποψη που ασχολούμαι με τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτό το οποίο με απασχολεί είναι να προσπαθήσω να βρω λύσεις ε, για να ξεπεράσω τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι χρήστες του Ιντερνετ. Also... Και επίσης να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι υπεύθυνε για το ίντερνετ και θα πρέπει τα δίκτυά τους να είναι πλήρως προσβάσιμα και ανοιχτά για όλους. Και θα δούμε αν εδώ υπάρχει μια κάποια δυνατότητα που να επιτρέψει τη συζήτηση και στα πλαίσια του ΠΟΕ. Ευχαριστώ κύριε Τίμανς. Η αντίδρασή σας και τα σχόλια σας δείχνουν ότι μπορούμε από κοινού να σκεφτούμε κάποια θέματα που θα μας επιτρέψουν να αναζητήσουμε λύσεις. Τα μέλη μπορούν να πάρουν το λόγο. και οι ομιλητές μεταξύ τους ε, είναι καλοδεχούμενοι να ανταλλάξουν απόψεις. Ας ε, ζητήσω λοιπόν πρώτον εάν τα μέλη μας θέλουν το λόγο. Η κυρία Αντρικίενε έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που ξεκίνησαν τη συζήτηση αυτή. Η συζήτηση αυτή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα, διότι το διαδίκτυο παίζει, όπως γνωρίζετε, έναν ρόλο πάρα πολύ σημαντικό στην ζωή όλων μας στην πολιτική και η σχέση μας γίνεται όλο ένα και πιο στενή με το ίντερνετ. Οπότε τι να πούμε τώρα, μετά από όλα αυτά που ξέρουμε από του εισηγητέ, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δώσουμε μάχη, γιατί να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στο Ιντερνετ και θα πρέπει όλο και περισσότερο να αυτό να είναι δυνατό και έχουμε και αυτές τις χώρες οι οποίες ελέγχουν όσο γίνεται, όλα για το, το διαδίκτυο το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ σημαντικό μέσο ώστε να υπάρχει κινητοποίηση και να υπάρχει ε, διαμαρτυρία και ταυτόχρονα έχουμε πάρα πολλές χώρες οι οποίες ε, ασκούν την λογοκρισία 60%. 60 χώρες, λέει, διορθώνει η ομιλήτρια, ασκούν τη λογοκρισία. Όπως είπε η κυρία Μοριών, έχουμε 72 blogs, στην bloggers, 72 bloggers στην Κίνα έχουν πάει φυλακή. Τρίων ετών λογοκρισία διακρίνουμε πολιτική για τον έλεγχο των πολιτικών ιδιών, για ε, λόγους ηθικής, για παιδική πορνογραφία, για τυχερά παιχνίδια, για ε, το, το κατέβασμα προστατευμένης πνευματικής ιδιοκτησίας. Βέβαια αυτά ισχύουν με διαφορές ανά χώρα και επίση και για εμπορικού λόγου γίνεται λογοκρισία, ούτω ώστε να υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Το πιο σημαντικό είναι να μπλοκαρίζονται κάποια site. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα που ακούστηκαν σήμερα από του ομιλητέ και ως μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου έχουμε όλες αυτές τις ε, συστάσεις να διατυπώσουμε και θα πρέπει οπωσδήποτε αυτό να το αντιμετωπίσουμε και να γίνουν ε, επαφές, διαβούλευση, διάλογος στο επίπεδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάτι άλλο πέραν αυτού είναι το τι θα γίνει μέσω του ΟΗΕ, μέσω του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ίσως είναι δυνατόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να περάσει ένα ψήφισμα σχετικά. Τρίτο σημείο τώρα είναι, θα μπορούσα να κάνουμε κάτι, είναι ο ΠΟΕ. Για πέστε μας. Τι μπορούμε να προτείνουμε προς ε, Συμβούλιο Κομισιόν. Τι πρωτοβουλίες μπορούν να αναλυφθούν. Ευχαριστώ. Συμφωνώ και εγώ, λέει πρόεδρος, με την ε, αντιπρόεδρο. Πέστε μας, τι μέτρα μπορούμε να περάσουμε, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Το κύριο Σομπιόλς έχει δει το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα πρώτα πρόεδρε θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους προσκεκλημένους μας που μας τίμησαν με την παρουσία τους απόψε γιατί πράγματι ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή η εισήγηση που μας έκαναν όλες αυτές οι απόψεις που ακούσαμε και κρίμα που έχουμε τόσο πολλές συνεδριάσεις στο Κοινοβούλιο και έτσι δεν μπόρεσαν να έρθουν περισσότεροι συνάδελφοι. Κρίμα, κρίμα, γιατί και αυτοί θα την εντυπωσιαζόντουσαν όπως και εμείς. Πρέπει να σας πω κάτι που κάποια στιγμή διάβασα από έναν ειδικό. Ειδικό στις νέες τεχνολογίες και στην κοινωνία της πληροφορίας τον Μανουέλ Καστέλς ο οποίος έγραψε πριν από μια δεκαετία νομίζω ένα τρίτο μου έργο στον αφορά την κοινωνία της πληροφορίας και θυμάμαι ότι στο Λονδίνο άκουσα τον Λούις Χάντον που έλεγε ότι είναι σαν τον Μάρξ ο Καστέλης. Αυτό το τρίτο μέρο της νέας πληροφορίας είναι κάτι σαν το κεφάλι του Μάρξ. Έλεγε ο Χούτον. Και για μένα πιο πολύ μετράει το, το έργο του ε, Καστέλης παρά του Μάρξ. Τέλος πάντων, το λέω για, για πλάκα. Επομένω είναι μεγάλη η αξία του. Και είχε πει ότι τα τελευταία χρόνια Δεκάδες κυβερνήσεων έχουν απευθυνθεί σε αυτόν και τον ρωτήσανε τι να κάνουν για να ελέγξουν το Ιντερνετ. Και πάντα απαντούσε είναι αδύνατο να ελέγξετε το Ιντερνετ. Μπορείτε να το ρυθμίσετε, αλλά δεν μπορείτε να το ελέγξετε. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες εθνικές ε, ιδιορυθμίες, κάποιες περιπτώσεις που έχουμε αυτό το φιλτράρισμα, έχουμε τη λογοκρισία, έχουμε τη χειραγώγηση που ουσιαστικά είναι προσβολές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών. Να είμαστε όμως αισιόδοξοι γιατί από πλευρά της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το Ιντερνετ είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό. Εγώ ζούσα 20 χρόνια υπό δικτατορία και καθόμαστε και βγάζαμε φυλάδια τυπώναν παράμε σε εφημερίδες για να τις μοιράσουμε. Επομένω, να, πόσο φανταστικό είναι τώρα το Ιντερνετ για έναν δημοκράτη, για έναν που παλεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα όμω. Υπάρχει ένας κίνδυνος. Δύο σπράφηγο για υποχρέωση μια άλλη συνεδρίαση, αλλά όμω δεν άκουσα να αναφέρεται ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα το οποίο με απασχολεί. Περισσότερο από το πιθανό έλεγχο ή την λογοκρισία του ίντερνετ είναι η απειλή από τον μεγάλο αδελφό ο κίνδυνος του να έχουμε ένα μονοπόλιο, ένα ολιγοπόλιο από αυτά τα μεγάλα, τα παγκόσμια μονοπόλια τα οποία να μπορέσουν να μπουν να αποκτήσουν πρόσβαση στην, στον ιδιωτικό βίο ε, να ελέγξουν δηλαδή τελικά αυτά τα προσωπικά δεδομένα του κόσμου. Πάνω σε αυτό θα να μου πούνε οι, οι δικοί μας τι πιστεύουν. Εγώ μπορώ τώρα να ανεβάσω μέσω του Google στο παγκόσμιο δίκτυο κάποια έγγραφά μου και δεν πειράζει γιατί δεν έχουμε κρύψει τίποτα αλλά είναι μια τέτοια τάση που διαφέρεται και που κάνει να διαφαίνεται ένα τέτοιο κίνδυνο για αυτή την ε, διάσταση που ξανήγεται. Επίσης, ο κ. Βάγκνερ δεν είναι τώρα πια εδώ, αλλά θα έπρεπε να συζητήσουμε και με αυτόν αυτά τα ζητήματα και να δούμε πώς θα αριστοποιήσουμε το δικό μας ρόλο σαν ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και στο κείμενο αυτό λέω ότι θα πρέπει να υπάρχει καλός συντονισμό μεταξύ των ε, θεσμικών οργάνων στην Ευρώπη. Γιατί όπως λέει εδώ, δεν έχουμε εξορθολογισμό αυτού, αυτού του, του συντονισμού του ρόλου μας. Άρα θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να έχουμε, τι, πού μπορούμε να προχωρήσουμε, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε πέρα από αυτή την κάπως διπλωματική διατύπωση του κ. Βάγκνερ. Ευχαριστώ πολύ. Προσθέσατε μια ουσιαστική διάσταση στη συζήτηση σχετικά με τα ιδιωτικά στοιχεία, την εμπιστευτικότητα των ιδιωτικών στοιχείων. Έχουμε άλλο ένα συνάδελφο που έχει ζητήσει το λόγο, ο David Μάρτιν. Όπως και η κυρία Αντρικίνε είναι μέλος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Ευχαριστώ, θα είμαι πολύ σύντομος. Θα ήθελα να επανέλθω στην παρουσίαση ε, την οποία έκαναν οι φιλοξενούμενοι μας και τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Για το Ιράν θα ήθελα να μας πείτε τι διαδικασίες έχετε θέσει σε λειτουργία στην επιχείρησή σας για να αποφύγετε ε, τέτοιου είδους καταστάσεις στο μέλλον. Ξέρω ότι δεν υπάρχουν 100% μέτρα τα οποία να αποτρέπουν τέτοιου είδους γεγονότα, αλλά ε, πώς μπορείτε να αποφύγετε να συνδέσετε το όνομά σας με υποκλοπές από πλευράς καθεστώτων ε, τα οποία θεωρούνται ύποπτα και υπάρχει δυνατότητα να θέσετε κάποια στάνταρτ έτσι ώστε όλες οι επιχειρήσεις να, είναι, να τα τηρούν και να λειτουργούν με συμβατό τρόπο. Υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας λοιπόν του συνόλου της βιομηχανίας παραγωγής τέτοιων συστημάτων. Ξέρετε ότι η Επιτροπή Εμπορίου ε, ασχολείται για διαφορετικούς λόγους βέβαια με το θέμα των ε, παραποιημένων εμπορικών σημάτων και προϊόντων. Ε, υπάρχουν πολλές μέθοδοι οι οποίες ακολουθούνται για την αντιμετώπιση της παραποίησης και ένας από τους τρόπους είναι να πάψει η διακίνηση αυτών των προϊόντων, η διακίνηση και η διαφήμιση τους μέσα από το διαδίκτυο. Δεν ξέρω τι μηχανισμός θα μπορούσε να υπάρχει για τον περιορισμό της κυκλοφορίας των προϊόντων αυτών μέσω του διαδικτύου. Ευχαριστώ κύριε Μάρτιν. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Δύο λεπτά παρακαλώ ο καθένας από τους ομιλητές που πήρε το λόγο προηγουμένως. Δεν έχω καλύτερη μέθοδο από το να προτείνω να ξεκινήσει ο κύριος Πούντεφατ, ο οποίος ε, συνέγραψε και την πρόταση τη γραπτή η οποία έχει γίνει. Κύριε Πούντεφατ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Μεγάλη ομοφωνία μεταξύ όλων όσων είμαστε εδώ σήμερα ότι όντως υπάρχει δυνατότητα τα, οι αξίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα να συμμορφωθούν με την δουλειά της Κομισιόν, του Κοινοβουλίου, των διαφόρων διεθνών οργανισμών, των εταιριών. Υπάρχουν, ε, υπάρχει κοινό τόπο λοιπόν, υπάρχουν και κάποια εμπόδια βεβαίω, υπάρχουν και νομικέ υποχρεώσει για τι διάφορε υπηρεσίε. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε, να προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, εφόσον θέλουμε να συνεργαζόμαστε σε ένα διεθνέ περιβάλλον. Και χαίρομαι για αυτό που είπε και ο κύριο Τίμα για τι συστάσει. Τώρα για τα θέματα της ε, ιδιωτικής σφαίρας. Είναι μεγάλη πρόκληση αυτό και αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο στην έκθεσή μας, αλλά δεν νομίζω ότι κάποια εταιρεία ή κυβέρνηση μπορεί να ελέγξει το ίντερνετ. Είναι κάτι που εξελίσσεται. Είναι ένα σύστημα που εξελίσσεται. Και είναι σημαντικό να έχουμε να μπουν αυτέ οι αρχέ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να είναι και σωστό ο τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί το ίντερνετ. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο που να απειλεί αυτό το σύστημα. Τώρα, το πρόβλημα θα υπάρξει αν δεν κοινοτοποιηθεί το κίνημα για τα ανθρώπινα δικαιώματα σημαντικά. Υπάρχουν μόνο κάποιοι που μπορούν ίσως ε, να προσπαθήσουν να περιορίσουν, να σταματήσουν την ανάπτυξη του ίντερνετ. είναι μια μυστική διαδικασία μα είπαν ε, αυτοί που υπεραμείνονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό προσπαθούμε να, μεταφέρουμε, να επιφέρουμε μεγαλύτερη διαφάνεια για να κινηθούν προ σωστή κατεύθυνση. Yeah, thank you very much. Uh, then, Mrs. Η κυρία Μοριό. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω κι εγώ για το ερώτημα για την άκτα. και μας μας ανησυχεί η, ε, να μας ανησυχούν οι δυνατότητες να περιοριστεί η ελεύθερη έκφραση στο διαδίκτυο. Δύο βασικά θέματα υπάρχουν στην έκθεση. Η ανάκληση της πρόσβασης ε, στην ε, πληροφόρηση. Θεωρούμε ότι είναι θεμελιώδες δικαίωμα η πρόσβαση στο ίντερνετ και επίσης αυτή η συνθήκη Ε, έχει οδηγήσει τους ενδιάμεσους να μετατρέπουν την, ε, ε, τα όσα ισχύουν σε πολιτική για, την, για, την, για τον έλεγχο των πρωτοκόλων για το ίντερνετ. Είναι πολύ σημαντικό να η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει, να φτάσει στον ΠΟΕ, να προσφύγει, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχουν εμπόδια στο ελεύθερο εμπόριο πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να παλύψουμε τα εμπόδια για την ελεύθερη έκφραση στο ίντερνετ. Βεβαίω οι επιχειρήσει είναι σημαντικό να συμβάλλουν, αλλά η λογοκρισία στο ίντερνετ είναι, και, είναι εμπόδιο και εμπορικό. Γιατί πώ μπορεί κανεί να διαφημίσει τι ε, εμπορικέ του δραστηριότητε, αν δεν υπάρχει ισόρροπη πρόσβαση σε ελεύθερη πληροφόρηση, πώ μπορεί να επενδύσει ε, Γι' αυτό μιλούμε. Δεν μιλούμε για την ε, παρεμπόδιση των ε, εμπορικών δραστηριοτήτων. Μιλούμε για την απάλληψη κάποιων εμποδίων. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί μόνο η, το freedom ε, of, η ελευθερία της έκφρασης μόνο από κάποιους λίγους Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει παγκόσμια συνεννόηση, ε, να συνεργαστούν η ΕΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πράξη για την ε, ελευθερία της έκφρασης ε, είναι μία από τις βασικές πράξεις. Είναι ένα νομοθετικό κείμενο που, δεν, που θα μπορούσε να αποτρέψει τις εταιρείες από το να περιορίζουν την ε, ελεύθερη έκφραση. Στην αρχή ε, κυρώθηκε μόνο από τη ΣΥΠΑ, μετά ξανάρχονται και κάποιες άλλες χώρες με το μέρος μου. Ε, Mr. French. Θέλουμε να το συζητήσουμε περισσότερο το θέμα αυτό. Υπάρχει ανάγκη για τέτοια για μια τέτοια συζήτηση, διαβούλευση. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα αναπάντητα. Θα ήθελα να απαντήσω σε μερικά. Καταρχήν, ποιες είναι οι δράσεις που, αναλάβαμε για να αξιολογήσουμε τα θέματα αυτά. Έχουμε έναν κατάλογο χωρών και προϊόντων που είναι επικίνδυνα σε ό,τι αφορά τι πωλήσει, όταν έχουμε θέματα που θεωρούμε ότι δεν μπορούν να λυθούν, όταν έχουμε προβλήματα, έχουμε μια διαδικασία που αναθεωρεί την όλη διαχείριση τη υπόθεση. Αναθεωρούμε τι πολιτικέ και τι πρακτικέ που έχουμε και η εμπειρία δείχνει ότι υπάρχει, πρέπει να υπάρξει σύσφυξη και να είναι πιο πρέπει να μάλλον να υπάρξει αυστηροποίηση και να είναι πιο διαφανή τα πράγματα. Το να δώσουμε μια απάντηση ναι ή όχι δεν είναι πάντα εύκολο. Και είναι μεγάλη πρόκληση επίσης όταν ως εταιρεία μας ε, ζητούν να δημιουργήσουμε δίκτυα σε χώρες που υπάρχουν σημαντικά θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ΟΗΕ μας έχει ζητήσει να δώσουμε δίκτυα σε χώρες που θα συμφωνούσατε όλοι ότι υπάρχουν σημαντικά θέματα, προβλήματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα. These cross Επίσης, ε, συμφωνώ ότι, ε, ότι έχουμε ξεκινήσει κάποιες ε, αρχικές δραστηριότητε. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Πρέπει να γίνουν περισσότερα, είναι σαφές. Και από την εταιρεία είμαστε στη δημοσιότητα συνέχεια. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία έχουν παρεξηγηθεί και Πρέπει να πω ότι αυτό δεν είναι κάτι που οι υπόλοιπε εταιρείε θα μας, ε, για το οποίο θα μας ακολουθήσουν. Θεωρώ ότι υπάρχουν ε, θέματα που πρέπει να τα λύσουμε ως ε, εταιρεία. Αλλά έχουμε λάβει και μια διαφορετική προσέγγιση. Ας πούμε στο Ιράν έχουμε περιορίσει τις δραστηριότητε μας. Δεν δίνουμε υπηρεσίες σε, τρίτες, σε τρίτους παρόχους στο Ιράν και οι ανταγωνιστές μας νομίζω ότι ε, έχουν, το έχουν υποστηρίξει. Εμείς υποθέσαμε ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση παρόλο που δεν είναι εύκολο να γίνει κατανοητή. Υπάρχουν πολλές αναφορές σε υψηλή τεχνολογία που χρησιμοποιείται και η πραγματικότητα είναι ότι σε πολλά δεν είναι υψηλή η τεχνολογία που χρησιμοποιείται. Δεν χρειάζεται δηλαδή υψηλή ε, τεχνολογία, δεν χρειάζεται σύστημα ή δίκτυο Alcatel ή Siemens ε, για να γίνει ο περιορισμός. Απλώς χρειάζεται γνώση και τεχνογνωσία. Μπορούμε ας πούμε, να δώσουμε ένα μόνιτορ που, ε, που μπορεί να υπάρχει και να υπάρχει όμως, να το έχουμε δώσει εμείς, αλλά να υπάρχει και από άλλους που θα μπορούσαν να το έχουν κάνει. Ναι, ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Ε, καλά θα ήταν να μπορούσαμε να συζητήσουμε περαιτέρω τα θέματα αυτά. Ο κύριος Χάντον τώρα ας πάρει το λόγο. Ε, thank you. When we took our moves in China, one, ε, some, some people... Όταν ασχοληθήκαμε με την Κίνα, μας είπαν ότι θα πρέπει να είσαστε αυστηροί λόγω του ότι έχετε και πάρα πολλοί αυστηρούς κανόνες για τη λειτουργία του Google στο διαδίκτυο. Να μου επιτρέψετε να σχολιάσω τώρα τις συστάσεις της κυρίας Αντρικίνα. Προφανώς θα εξετάσουμε την δυνατότητα συζήτησης του θέματος των ΠΟΕ. Αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον για εμπορικούς εταίρους όπως εμείς. Το GNI ακριβώς όμως υπάρχει για να διαμορφώσει αυτόν τον ε, τρόπο θα έλεγα συμπεριφοράς όλων των εμπλεκομένων επιχειρήσεων. Είναι κάτι το οποίο υπέγραψαν τρεις μηχανές αναζήτησης από τις ανωμένες Πολιτείες, αλλά μετά ε, ε, συνήψαν συμφωνία και άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες όμως τελικά στο τέλος μάλλον δεν πήραν μέρος στην προσπάθεια. Ο έλεγχος. Ο έλεγχος είναι θα έλεγα αυτή η λέξη που έχει σημασία στην κοινωνία γνώσης του 21ου αιώνα. Δεν μπορεί κανείς ε, να σταματήσει την καινοτομία, την επαναστατική καινοτομία και την ελεύθερη έκφραση στο διαδίκτυο. Αυτά είναι σαφή. Το θέμα είναι όταν κάτι ξεφύγει μπορεί να περιοριστεί εκ των υστέρων μήπως ε, υπάρχει δυνατότητα ε, να νομοθετήσετε με διαφορετικό τρόπο έτσι ώστε να προστατευτούν τα ιδιωτικά δεδομένα. Οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα στα δεδομένα τα οποία καταθέτουν ή παίρνουν από το διαδίκτυο. Η κυρία Μοριό είπε ότι το βασικό πρόβλημα από πλευράς μας είναι η μεταφορά της ευθύνης στους ενδιάμεσους. Αυτοί οι οποίοι δημιουργούν τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται για τηλεπικοινωνίες θεωρούνται υπεύθυνοι για αυτά τα οποία βάζονται πάνω σε αυτές τις πλατφόρμες. Αντίθετα, οι πλατφόρμες αυτές είναι ελεύθερες και δεν μπορούμε εμείς να γίνουμε αστυνομικοί. Και δεν μπορούμε να δημιουργούμε συστήματα τα οποία να είναι κλειστά και να ελέγχονται εύκολα τελικά από τις κυβερνήσεις. Ευχαριστώ κύριε Χάμπτον. Εγώ δεν γνώριζα το Global Network Initiative, το GNI, και θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή και των ευρωπαϊκών εταιριών στην πρωτοβουλία αυτή. Όπως είπε και ο David Martin, μερικές φορές οι ε, συμφωνίες αυτές σε εθελοντική βάση είναι αφετηρία ίσως ε, για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας η οποία να λειτουργήσει πραγματικά ισότιμα. Ο κύριος Τσούο. Ε, χαίρομαι που τέθηκε το θέμα των ιδιωτικών στοιχείων, ιδιωτικών δεδομένων και των πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτά είναι θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν ε, γιατί συνδέονται και με την οικονομική άποψη. Σε επίπεδο τεχνικό από τις εμπειρίες που έχουμε τα τελευταία χρόνια Πολλά από τα θέματα αυτά αφορούν την ανάπτυξη λογιστικού είτε για παραγωγή είτε για έρευνα. Είναι στην ουσία ένα παιχνίδι της γάτας και του ποντικού. Νομίζω μιας και αναζητούμε μια σωστή λύση προστασίας των ιδιωτικών δεδομένων και της πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι θέμα παιδείας θα έλεγα για να αντιμετωπίσει ο κόσμος με σωστό τρόπο το πρόβλημα το οποίο έχουμε. Και όταν η κοινωνία το κατανοήσει τότε θα λυθεί το πρόβλημα. Θα ήθελα να πω επίσης ότι η πιο φρικτές επιθέσεις στο ίντερνετ σε αυτή τη φάση ξεπερνούν τα προβλήματα της πνευματικής ιδιοκτησίας ε, και της, των ιδιωτικών δεδομένων. Αφορούν θέματα ε, εθνικών, ε, σαν παράδειγμα, προβλημάτων εθνικής ασφαλείας. Υφιστάμεθα στην Κίνα επιθέσεις τα αμυντικά μας συστήματα. Το ίδιο γίνεται και με ηλεκτρονικές επιθέσεις από από δίκτυα όπως το GhostNet, όπως λέγεται, ε, στις Ηνωμένε Πολιτείες, στο Κογκρέσο. Στις Ηνωμένε Πολιτείες θεωρείται ότι ο έλεγχος του ίντερνετ είναι κάτι το καλό βέβαια για την κρατούσα τάξη. Και αυτό δεν ξέρω αν είναι μια σωστή λύση. Αν δεν λυθεί λοιπόν το πρόβλημα της λογοκρισίας στην Κίνα και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υποστηρίξει την ελεύθερη κυκλοφορία ιδεών στο διαδίκτυο, τότε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με την Κίνα ε, θα κρατήσει πάρα πολλά χρόνια και θα βρεθεί εκτός ελέγχου. και υπάρχει πάντα το πρόβλημα όπως είπα των, της, του βίαιου χαρακτήρα των επιθέσεων ε, στο διαδίκτυο και αυτό θα αφισβητήσει ε, την δυνατότητα πρόσβασης στην ελεύθερη επικοινωνία όλων των κλειστών κοινωνιών. Yes, it's on. Α, αναμένω το μικρόφωνο. Ναι, δεν είστε μόνος που πιστεύει ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε προς το, προς το του, του ΠΟΕ. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι αυτονόητο, οπότε πάλι καλά. Να, και εγώ να σας πω σε σχέση με τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν ποια είναι η σχέση εμπορίου και ανθρωπινών δικαιωμάτων που φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό τα θέματα που συζητήθηκαν. Και αυτές οι συμφωνίες εμπορίου. Μάλλον απεσιόδοξο είμαι. Δεν έχουμε απόδειξη ότι είναι δυνατόν να αποδώσουν ρήτρα των δικαιωμάτων. Αν γινόταν έτσι, δεν θα γινόντουσαν καν συμφωνίε. Ο κόσμος θέλει απλώ να κλείσει τις συμφωνίε. Βρισκόμαστε σε έναν κόσμο που βασιλεύει ο ανταγωνισμός. Και είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνούμε ότι συνεχώ, αγοράζουμε αγαθά, υπηρεσίε, εμπορεύματα, αναδεχόμεθα από εκείνες τις οικονομίες που, που, που, που συζητούμε τους εργαζόμενους και αν βάλουμε τέτοιε ρήτρε τότε θα κάνουμε τις συμφωνίες σχετικές. Δεν θα δώσω την απάντηση, αλλά υπάρχουν διαφορές συνταγματικέ, νομικές μεταξύ ημών και εκείνων και τέτοιου είδου ε, ανοίγματα είναι δυνατόν να αποτελέσουν μπούμεραν για εναντίον μας. Γιατί κάποιε χώρε έχουν τελείω διαφορετική άποψη όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία. Οπότε με το επιχείρημά μα θα μα απαντήσουμε ένα αντεπιχείρημα. Και ε, το σχετικό με την ε, ευθύνη είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι έχει να κάνει με κάποιον μη κρατικό παράγοντα οπότε κάποια δεσμικά όργανα όπως ε, εσείς δεν προστατεύει τις επιχειρήσεις βιομηχανίας γιατί αφήνεται να αποφασίσει άλλος για τις επιχείρησεις σας. Για δε το Ιράν έχουμε ένα δίλημα. Κατά πώς να δούμε το ίδιο υλικό, με την ίδια υποδομή, να έχουμε Twitter και ταυτόχρονα να έχουμε την ελευθερία λόγου. Μια που το ίδιο υλικό μπορεί και να διευκολύνει το Twitter, για την μετάδοση πληροφορία και να, και να την περιορίσει. Γι' αυτό και εγώ είμαι κάθετα εναντίον αυτή τη ιδέα όπως προείπατε. Δεν έχει νόημα αν μόνο μια-δυο χώρε προσυπογράψουν αυτή την συμφωνία για την ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών. Θυμάστε το πείρημα ότι αν δεν κάνουμε εμείς ε, το άνοιγμα θα το κάνει κάποιος άλλος. Τέλος πάντων αυτά είναι προσωπικές μου σκέψεις αλλά θεωρώ ότι έτσι η σύνδεσή μου είναι ήσυχη και είμαι ήσυχο. Αισθάνομαι ασφαλέστερος. Επομένως, προσοχή, τι γίνεται με την ευθύνη, την νομική ευθύνη, ε, όταν την αναθέτουμε σε κάποιον εκτός κρατικής δομής. Όχι, επίση έχουμε κάνει πάρα πολλά τόσο ώστε να αποτρέψουμε τι κρυφέ διαπραγματεύσει με κάποιε χώρε σε σχέση με το ΑΚΤΑ. Ο κύριο Τίμαν θέλει να υποβάλει μια σύντομη παρατήρηση και κατόπιν θα ολοκληρώσουμε αυτή, την ακρόαση τόσο ο Τίμαν. Και εγώ θα ήθελα να διαβιώσω εδώ τον παρακαθήμενο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι αναφανδόν υπέρ τη ελευθερία τη έκφραση και τη ελευθερία των ε, ε, μέσων επικοινωνίας και υπέρ της ελευθερίας του Ιντερνετ. Όλα αυτά τα θέματα τα έχουμε θίξει με Αίγυπτο, την Ισία, Κίνα και, και με άλλες χώρες. Βέβαια το θέμα είναι αρκούν αυτά για να τους πείσουμε να αλλάξουν στάση. Το είπα και προηγουμένω. ότι θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει όσον αφορά την εταιρική ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δύο σχετικές μελέτες εκπονήσει και θα πρέπει να το κοιτάξουμε. Τώρα, ε, αφού θα κλείσω εγώ, την ακρόαση πρέπει να σας πω ότι αν εγώ είχα την εκτελεστική εξουσία που δεν την έχω, είμαστε εδώ κοινοβούλιο, δεν είμαστε εκτελεστικό όργανο, θα έλεγα ότι εσείς μπορείτε να συγκροτήσετε μια, μια, μια ομάδα εργασία, ώστε να βοηθήσετε τους νομοθέτες και έτσι να προχωρήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν μπορώ και έτσι δεν το κάνω. Πάντως, σαν συμπέρασμα, κατόπιν των όσων είπατε και προτείνατε, είναι ότι κατά κάποιο τρόπο έτσι αρχίζουμε να ρίχνουμε φως σε έναν πολύ ενδιαφέροντα τομέα που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ίσως τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, λίγο μας μπερδεύουν, αλλά νομίζω ότι διανοίγεται μια δυνατότητα παρέμβασης. Εμείς δεν θα σταματήσουμε πάντως αυτό το θέμα να το προωθούμε και προς την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντως θα έχουμε μια εκδήλωση με τους φίλους του Freedom House. Είστε προσκεκλημένοι ακόμα και στο κτίριο. Με τους φίλους επίσης από Βορειοαφρική, από αραβικές χώρες και αν θέλετε να τα πούμε πιο χαλαρά είστε πρόσδεκτοι. Οπότε σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η ακρόασή μας και να δούμε το τελευταίο μας ε, θέμα για σήμερα. Είπαμε ότι ξεκίνησαμε με την ε, σύντομη συνέντευξη τύπου σε συνεργασία με το Freedom House και με τους δύο ομιλητές οι οποίοι είναι προσκεκλημένοι για σήμερα. Πρόκειται για τις μεταρρυθμίσεις στον αραβικό κόσμο. And ε, Freedom House is... Η Freedom House είναι μια μη κυβερνητική αμερικανική οργάνωση. Yeah. Συνεργαζόμαστε τακτικά μαζί τους και όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται είναι ανεξάρτητος εποπτικός οργανισμός σε σχέση με την ελευθερία σε όλο τον κόσμο γιατί προωθεί τις δημοκρατικές ε, αλλαγές ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα συγκροτήθηκε το 1941 έχουμε εδώ πέρα τρία και εκλεκτά στελέχη του φορέα αυτού και θα μας μιλήσει για αυτές τις αλλαγές τον κύριο Ανουάρ Σαντάτ από την Αίγυπτο. Έχουμε επίσης και τον Φοντίλ Μπουμαλά από την Αλγερία. Επίσης τον δόκτωρα Μουνίρα Φάκρο από τον Μπαχρέιν. So uh, Επομένως, για ένα δεκάλεπτο δώσουμε τώρα το λόγο και θα είμαι πάρα πολύ αυστηρή με το χρονικό όριο της αγόρασης, διότι θα πρέπει να υπάρχει περιθώριο να συζητήσουμε μετά. Δέκα λεπτά επομένως ο καθένας από τους αγορητές και πρώτος, αλλά ας λάβει το λόγο ο κύριος Ανουάρ Σαντάτ για να με ενημερώσει όσον αφορά το τι έγινε μετά από ε, αυτή την έκτακτη νομοθεσία κατάσταση ανάγκης που επικρίθηκε τόσο πολύ στην Αίγυπτο. Μας πει λοιπόν ο κύριος Σαντάτ τι γίνεται όσον αφορά τα μέτρα καταστολής στην ε, Αίγυπτο σε σχέση και με τις ε, εκλογές που θα γίνουν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε της Υποεπιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αγαπητά μέλη της Επιτροπής και προσκεκλημένοι όπως τα γνωρίζετε όλοι πριν από δέκα μέρες παρατάθηκε η διάρκεια της κατάστασης πολιορκίας και όπως ξέρετε αυτό το περιμέναμε παρά το ότι ο Πρόεδρος κατά την προεκλογική στρατεία είχε υποσχεθεί το 2005 δηλαδή ότι θα έθετε τέλος. σε αυτή την κατάσταση πολιτικής που κρατεί 29 χρόνια, αλλά όμως δεν έγινε τίποτα. Από το 2005 έγινε παράταση διετής, άλλη μια παράταση διετής και θεωρώ ότι θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση έως ότου γίνουν οι εκλογές τον Νοέμβριο τότε έτους και επίσης θα έχουμε και τις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν περί τα τέλη του 2011. Βέβαια υπάρχουν κάποια επιχειρήματα και λένε ότι ο νόμος περί καταστάσεως πολιορκίας ε, χρησιμοποιείται μόνο κατά των ναρκωτικών και κατά της τρομοκρατίας. Όμως κατά αυτά τα 29 χρόνια μάλλον συνεχίστηκε οι εμπόροι ναρκωτικών. Υπάρχουν ναρκωτικά παντού. Και έχουμε και κάποιες τρομοκρατικές συνέργειες στην ε, Αίγυπτο. όμως δεν ωφέλησε στο να φρενάρουμε κάποια αυτά τα φαινόμενα. Όμως αυτό ήταν δικαιολογία, αύξηση του κύρους, της εξουσίας, δυνατότητες να ελέγξουν την πολιτική ζωή στην Αίγυπτο. Και όπως προείπα, παρά τις προεδρικές υποσχέσεις της προεκλογικής εκστρατείας, δεν συνέβη τίποτα. Είδατε χθε, παρετήθηκε ο Ιαπωνέζος Πρωθυπουργός μόνο και μόνο γιατί είχε δώσει την υπόσχεση ότι θα έδιωχνε μια, μια βάση Αμερικάνη στην Οκινάβα νομίζω. Δεν το έκανε και παρετήθηκε. Όμως αυτά γίνονται στην Ιαπωνία. Οπότε, βλέπετε. Έλεγχος σημαίνει αυτή η νομοθεσία. Κατά των ακτιβιστών χρησιμοποιείται για τις εκλογές, ε, ε, πρόβλημα ε, του συναθρίζεστε, πρόβλημα όσον αυτό το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε, τέλος πάντων και έχουμε στατοδικεία αντί για τακτικά δικαστήρια. Όλο ειδικά δικαστήρια για τις παραδιάσεις αυτής της νομοθεσίας. Και αν παρακολουθήσεις και λήξεις στην, ε, στην, στην Αίγυπτο έχουμε ένα σωρό συλλαλητήρια από όλα τα κομμάτια της κοινωνίας. Δάσκαλους, γιατρούς, ε, όλοι παρά στην Αίγυπτο. Και είχαμε μια δημοσίευση, ένα... Α, συγγνώμη, είχαμε το άρθρο 3 παράγραφος 1 που προβλέπει ο νόμος για κατάσταση της ανάγκης που λέει ότι προσθέτεται η δυνατότητα στην κυβέρνηση να κάνει ό,τι θέλει οποτεδήποτε. Και δεν υπάρχει ένδικο μέσο κατά μια τέτοια απόφαση και αυτό και έγινε. Ετελέστησαν οι εκλογέ, η Σούρα, αυτό το συμβούλιο χθε, συγκροτήθηκε, συνήρθε και είχαμε πάλι τα ίδια εκλογέ. καταγγελίες της ε, αντιπολίτευση ακόμα και από την ε, μουσουλμανική αδελφότητα. Τους κλειδώσαν. Τους περιορίσανε, τους δίρανε. Και όλα αυτά δυνάμει της νομοθεσίας αυτής για κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κάποιοι ασιάτες, κάποιοι ψηφοφόροι που δεν τους αφήσαμε να πάνε να ψηφίσουν. Χτες μόλις γίνανε όλα αυτά. Και το πρόβλημα είναι ότι έχουμε τώρα μια εκλογική επιτροπή που εποπτεύει. Όμως και αυτή είναι δοτή. Τους ορίζει, τους διορίζει ο πρόεδρος. Ακριβώς όπως έχουμε και το Εθνικό Σύμβολο των Ανθρώπινα Δικαιώματα που και αυτή υποτίθεται είναι ανεξάρτητη αλλά και αυτοί διορίζονται και έχουν κάποια όρια στις δυνατότητες τους που δεν μπορούν να τα υπερβούν. Να, είναι πάρα πολύ καλή η κυβέρνηση σε αυτό. Να συγκροτεί τέτοια συμβούλια, εθνικά συμβούλια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και λοιπά. Όλα αυτά τα συμβούλια τα φτιάχνουν για να συμμορφωθούν προς τα διεθνή πρότυπα. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά τελικά όλα αυτά τα συμβούλια δεν είναι ανεξάρτητα. Όμως, μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έπρεπε να πιέσουμε να προβάλλουμε το ότι κάτι γίνεται αλλά δεν βγαίνει όλη η αλήθεια γιατί ουσιαστικά είναι κομμάτι της κυβέρνησης και αυτά τα συμβούλια Επομένως η κυβέρνηση και το κυβερνόν κόμμα είναι πάρα πολύ καλή στο να επιλέγουν τους εκπροσώπους. Αυτούς που έρχονται εδώ συναντούν και μιλούν με τη δική σας με επιτροπή ή με άλλους ε, εκπροσώπους της Ένωσης και δικαιολογούν ό,τι γίνεται λέγοντας ότι να, η Αίγυπτος περικλείεται από τόσους εχθρούς, έχουμε τη Γάζα, έχουμε τη Χαμάς, ε, κοντά μας είναι στη γειτονιά μας και ο πόλεμος του Ιράκ. βρίσκουν ένα σωρό δικαιολογίε. Και λένε, επομένω είναι έκτακτη κατάσταση που, που επιβάλλει ε, ε νομοθεσία και τι για την εθνική ασφάλεια. Ο όμως θα πρέπει να βρεθεί κάποιο είδου εξισορρόπηση μεταξύ αυτονών, της κοινωνίας των πολιτών και των ανεξαρτήτων βουλευτών. Των βουλευτών της αντιπολίτευσης τέλος πάντων. Θα πρέπει να κάτσουν και να τα συζητήσουν στη βάση του διαλόγου ακόμα και με τους ε, μουσουλμάνους αδελφότητας. Δεν μπορούμε να τους αγνοούμε γιατί είναι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Να τους ακούσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι τους στηρίζουμε, ότι συμφωνούμε μαζί τους, αλλά θα πρέπει να δοθεί αυτή η ευκαιρία. Ευκαιρία, όπως ώστε να δούμε τι θέλει ο λαός. Γι' αυτό σας λέω. Και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ εγώ κύριε Σαντάμ που μας τα ε, εξηγήσατε όλα αυτά την τόσο κρίσιμη κατάσταση της χώρας σας. Ο κύριος Μπουμάλα από την Αλγερία τώρα. Βρεθήκαμε και στην ε, συνέδευξη τύπου σήμερα το μεσημέρι. Θα μιλήσετε για την ελευθερία της έκφρασης μεταξύ άλλων στην Αλγερία. Έχετε το λόγο λοιπόν. Madame Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, θα θέλαμε μέσα από αυτή την παρουσίαση να ακουστούμε στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης μας και στα πλαίσια των στοιχείων τα οποία έχουμε συλλέξει επιτόπου και ε, δεν νομίζω ότι θα πρόκειται για μία απλή παρουσίαση στα πλαίσια μιας παραδοσιακής ακρόασης. Να εκφέρουμε επίσης και κάποιες διαπιστώσεις, κάποιες εικόνες της πραγματικότητας σχετικές με τα σημεία τα οποία σε πολιτικό, θεσμικό, νομικό και λειτουργικό τρόπο λειτουργούν σαν εμπόδια είναι εμπόδια τα οποία γενικότερα βάζουν την κοινωνία και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους δημοσιογράφους ιδιαίτερα σε πολύ δύσκολη θέση. Η Αλγερία θα έλεγα γνώρισε ένα πέρασμα στη δημοκρατία το οποίο αρχικά ήταν αξιοπρεπές. Υπήρξε το πρόβλημα με την θρησκευτικά φανατική αντιπολίτευση. Και αυτό προκάλεσε σε υπερβολές και οδήγησε σε μια κατάσταση συμφιλίωσης ανάμεσα στους δύο εταίρους της κρίσης. Αυτούς που προκάλεσαν δηλαδή την κρίση. Και η κοινωνία τελικά ένιωσε ότι έχει παγιδευτεί και αυτήν την κοινωνία εκπροσωπούμε και εμείς σήμερα την κοινωνία η οποία αν θέλετε τελικά κλήθηκε να πληρώσει το λογαριασμό. Πραγματικά ένα λογαριασμό ο οποίος δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα σε αρκετά σημεία. Η Αλγερία στις αρχές της δεκαετίας του 80 ήταν υπόδειγμα σε επίπεδο ελευθερίας τύπου και δημιουργίας ε, μέσων ενημέρωσης. Εδώ και δέκα χρόνια υπαναχωρεί συστηματικά σε σχέση με την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία δημιουργίας ε, ίδρυσης εφημερίδων και μια συνεχούς παρεμβατικότητα της κυβέρνησης και των δυνάμεων ασφαλείας στα πλαίσια της άσκησης των δικαιωμάτων ε, του λειτουργήματος της ενημέρωσης. υπάρχει πάντα η αίτηση αδειοδότησης ε, για να ξεκινήσει κανείς οποιαδήποτε δημοσίευση στην Αλγερία, είτε πρόκειται για ημερήσια εφημερίδα είτε για μηνιαίο περιοδικό. Υπάρχει μια απόπειρα ελέγχου των πάντων και των μέσων, νέων μέσων ενημέρωσης μέσω του διαδικτύου. Γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί σύντομα ε, να καταθέσει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για να μπλοκάρει ουσιαστικά ε, την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα του πληθυσμού της Αλγερίας. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία επίσης δεν συζητάει το καθεστώς στην Αλγερία ή τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα και στον ιδιωτικό τομέα που θα μπορούσαν να εκφράσουν και τις απόψεις της πολιτικής αντιπολίτευσης. Η πολιτική αντιπολίτευση αντιμετωπίζει και αυτή τρομερά προβλήματα γιατί δεν έχει πρόσβαση στις εφημερίδες και στον δημόσιο γενικά χώρο, σε κάθε ε, είδος δηλαδή συγκέντρωση και διαδήλωση που δεν θα περάσει από αδειοδότηση των κεντρικών υπηρεσιών. Σε επίπεδο ποινικού δικαίου υπάρχει επίσης ένας νόμος ο οποίος χρησιμοποιείται σαν σπάθη του Δαμοκλέους επί της κεφαλής όλων των δημοσιογράφων και διανοουμένων που θα ήθελαν να εκφραστούν. Αυτός ο νόμος αφορά την, τον περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης και της φυλάκισης των δημοσιογράφων. Ε, μια χώρα η οποία αντιμετώπισε τρομερά προβλήματα στο παρελθόν και η οποία όμως διώκει τους δημοσιογράφους σήμερα, διώκει τις εφημερίδες, ε, τους υπεύθυνου σύνταξη. Πρόκειται για μια θα έλεγα επιστροφή στο παρελθόν η οποία δεν είναι καθόλου ε, σωστή και δεν υπερασπίζεται σε καμία περίπτωση τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα, θεσμικά περισσότερο, η κατηγορηματική άρνηση να προσφέρουν σε όσους παρεμβαίνουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες και την ηλεκτρονική ενημέρωση. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα εμπασπέπτω στον τομέα της ενημέρωσης, υπάρχουν προβλήματα ουσίας, διαφθοράς, βασανιστήριων κτλ. Τα πράγματα πηγαίνουν δυστυχώς ανάποδα και φύγονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της Αλγερίας. Το δικαίωμα οργάνωσης, όπως είπα, το δικαίωμα συγκέντρωσης, το δικαίωμα το να διαφωνεί, εν πάση περιπτώσει, κανείς με τις πράξεις της εξουσίας. Το υπάρχει και μια συνενοχή, αν θέλετε, ανάμεσα στους εταίρους της σημερινή εξουσίας, που κλείνουν όλες τις δυνατότητες έκφρασης και για τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τα πολιτικά κόμματα. Θα θέλαμε λοιπόν να κάθε εταιρική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αλγερία να περνάει μέσα από το θέμα του σεβασμού της ελευθερίας έκφρασης της κοινωνίας της Αλγερίας. ένα ανεξάρτητο ευρωμεσογειακό ή ευρωαραβικό ε, παρατηρητήριο θα ήταν ένας καλός τρόπος ε, παρακολούθησης καταστάσεων παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελευθερίας έκφρασης και άσκησης βασανιστήριων. Τέλος, είναι απαραίτητο για μας σήμερα και είμαστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπείτε τους λαούς της Ευρώπης. Ήρθαμε εδώ για να ακούσουμε τους λαούς της Ευρώπης και όχι τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, γιατί αυτές οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις τελικά ενισχύουν τα ολοκληρωτικά καθεστώτα στην περιοχή μας και στη Βόρεια Αφρική. Νομιμοποιούν τα καθεστώτα αυτά για πάρα πολλούς λόγους Υπάρχει το θέμα της ε, καταπολέμησης της τρομοκρατίας στην περιοχή που χρησιμοποιείται για πίεση της κοινωνίας. Από το 1992 ξέρετε ότι η Αλγερία ζει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην ουσία στερεί όλες τις δυνατότητες ελευθερίας και τα βάζει όλα υπό τον έλεγχο του καθεστώτος και των δυνάμεων ασφαλείας ακόμα και τους βουλευτές ένα καθεστώς έκτακτης ανάγκης λοιπόν το οποίο μας εμποδίζει να δράσουμε ελεύθερα. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στην ουσία δίνει δυνατότητες ενίσχυσης της παρουσίας των καθεστώτων αυτών λόγω της καταπολέμησης της ε, τρομοκρατίας και λόγω και της προστασίας των οικονομικών εταίρων. Η προστασία λοιπόν των οικονομικών συμφερόντων των ευρωπαϊκών χωρών συνιστά για μας μια έμεση συνενοχή των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων που απαγορεύει τις διαδικασίες αλλαγής και μετάβασης και θέτει σε αμφισβήτηση τις βασικές αξίες της δυτικής δημοκρατίας και σε επίπεδο αρχών και σε επίπεδο δράσεων των θεσμών και των οργάνων τους. Αυτό που έχει σημασία για μας σαν κοινωνία των πολιτών είναι να δημιουργήσουμε και να ενισχύσουμε τα κοινωνικά δίκτυα ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της κοινωνίας των πολιτών, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους δημοσιογράφους, όπως επίσης και της ε, πολιτικής πρακτικής ε, παιδαγωγικά θα έλεγα και για την πολιτική τάξη και για τους δημοσιογράφους και για τους διανοουμένους και για όσους όλους εν πάση περιπτώσει παραμβαίνουν σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο έντυπων μέσων ενημέρωσης για να προωθήσουν την δημοκρατία και τον εκδημοκρατισμό. Παίρνουμε το λόγο λοιπόν όχι να σα ζητήσουμε να αναλάβετε εσεί τι δικέ μα ευθύνε, γιατί η αλλαγή δεν θα προέλθει από την Ευρώπη ή από τι Ηνωμένε Πολιτείε, θα προέλθει μέσα από τι χώρε αυτέ, μέσω των τοπικών πρωταγωνιστών και εταίρων αρκεί να υπάρχει όμως μια εταιρική σχέση σε επίπεδο κοινών δράσεων, κοινών αξιών και μια συνεργασία ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών και μέσω των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών της Ευρώπης στη συγκεκριμένη περίπτωση τους οποίους σήμερα έχουμε την τιμή να ενημερώνουμε γιατί εσείς επηρεάζετε την κοινή γνώμη και γι' αυτό υπολογίζουμε στη βοήθειά σας. Σας ευχαριστώ που εκφράζετε την εμπιστοσύνη σας στο Κοινοβούλιο. Ελπίζω να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας να καλωσορίσω τώρα τον ε, γιο του κυρίου Χαϊτάμ Αλμαλέκ, υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καλωσορίσατε και εκ μέρους του Κοινοβουλίου σας καλωσορίζω Θέλετε, έχετε ζητήσει από την κυβέρνηση της Συρίας να απελευθερώσει τον πατέρα σας που βρίσκεται. Είναι φυλακισμένος με, για λάθος λόγους, ακριβώς μόνο και μόνο επειδή α, υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα θα περάσουμε στα θέματα των δικαιωμάτων των γυναικών και της πολιτικής συμμετοχής. Η κυρία Μονίρα Φάχρο είναι εδώ, η οποία θα μας αναφέρει. Θα μας κάνει την παρουσίαση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κυρία Πάρα έχει το λόγο. Τα θέματα των δικαιωμάτων των γυναικών έχουν λάβει μεγάλη σημασία, ειδικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, συγκεκριμένα από το 1995 με, την, ε, με τις συστάσεις ε, της ε, Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις γυναίκες στο Πεκίνο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το ο οικογενειακό δίκαιο έχει, είναι πολύ αναπτυγμένο στην Τινησία και το Μαρόκο. Ενώ οι υπόλοιπες αραβικές χώρες έχουν πολύ πιο συντηρητικό δίκαιο. Η Σαουδική Αραβία δεν έχει οικογενειακό δίκαιο αναφέρεται κατευθείαν στον κώδικα της Σαρία για τέτοια θέματα. Εδώ θα ήθελα να πω, να σας αναφέρω την μελέτη που έγινε από το Freedom House, μια πολύ σημαντική μελέτη, ένα πολύ σημαντικό project που υποστηρίζει εθνικές, την εθνική και διεθνή ευαισθητοποίηση για τις γυναίκες στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, ειδικά στον, στις χώρες του κόλπου, όπου οι γυναίκες υποφέρουν από την έλλειψη ε, νομοθεσίας και την διακριτική μεταχείριση. Το project αυτό δημιούργησε μεγάλη ευαισθητοποίηση μεταξύ και ανδρών και γυναικών, αλλά και των χαρασόντων την πολιτική. Προσπαθήσαμε λοιπόν να βασιστούμε σε αυτές τις πληροφορίες. Παρόλο που η έρευνα έδειξε ότι υπάρχουν ουσιώδεις ε, δυσκολίες και ελλείψεις ε, για τα δικαιώματα των γυναικών στις αραβικέ χώρες περιλαμβάνει και τη μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί την τελευταία δεκαετία για την κατάσταση που επικρατεί σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των γυναικών. Τώρα, να περάσω στο άλλο θέμα, το οποίο επίσης θεωρώ ότι είναι σημαντικό, το θέμα των πολιτικών μεταρρυθμίσεων στον αραβικό κόσμο. Τρεις αραβικές χώρες θα διεξάγουν εκλογέ φέτος. Η όλη διαδικασία των εκλογών σε όλες τις αραβικές χώρες πρέπει να μεταρρυθμιστεί σύμφωνα και με τις ανάγκες που έχει κάθε χώρα. Ένα παράδειγμα. Η δική μου χώρα, το Μπαχρέιν, θα διεξάγει εκλογές τον ε, Οκτώβρη του τρέχοντος. Το κοινοβούλιο αποτελείται από 80 βουλευτές. 40 διορίζονται και 40 εκλέγονται. Το Μπαχρέιν χωρίζεται σε 40 περιφέρειες. Αυτές οι περιφέρειες είναι χωρισμένες, κάποιες έχουν 16.000 ε, ε, ψηφοφόρους, κάποιες έχουν 600. Το ε, Μπαχρέιν απέρριψε όλους τους διεθνείς παρατηρητές. Η Επιτροπή που, ελέγχει, που παρακολουθεί τις εκλογές δεν είναι ανεξάρτητη, είναι διορισμένη από την κυβέρνηση. Λόγω λοιπόν όλων αυτών, Έγινε μεγάλη απάτη και ζητούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας βοηθήσει ώστε να μπορέσουμε να διεξάγουμε σωστά τις εκλογές. Επίσης, για τα θέματα της, ε, των δικαιωμάτων των γυναικών, ε, μεταρρύθμιση της νομοθεσίας ε, για το οικογενειακό δίκαιο, για τα θέματα βία στο, στο σπίτι και επίσης να ζητήσουμε την ε, δημιουργία μηχανισμών ε, ώστε να διευκολύνουμε τις γυναίκες να συμμετέχουν στην όλη διαδικασία λήψης αποφάσεων με ίσες ευκαιρίες. Αυτό για τις γυναίκες. Τώρα, για τις εκλογές θα θέλαμε να συζητήσουμε να μας βοηθήσετε να δημιουργήσουμε μια επίσημη εταιρική σχέση με τις χώρες εταίρους στον τομέα της παρακολούθησης, της κατάρτισης και της, του καθορισμού των προτύπων για την διεξαγωγή των εκλογών. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα θέλαμε να ζητήσει από τις, από τις χώρες εταίρους να εξασφαλίσουν ότι οι εκλογές θα γίνονται υπό την εποπτεία ανεξάρτητων επιτροπών, εκλογικών επιτροπών. Αυτό ζητούμε από εσάς και αν είναι δυνατόν θα θέλαμε μια απάντηση από εσάς. Αν έχετε ερωτήματα, ευχαριστώ να απαντήσουμε. Thank you very much, Mr. Εμείς σας ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος. Πολύ διατυπώσατε για προτάσεις σε σχέση με το τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να σας βοηθήσει το έργο σας. Και βέβαια πρέπει να ευχαριστήσουμε το Freedom House που σα βοήθησε να έρθετε εδώ, ο καθένας από τη χώρα του και εμεί ε, θα πρέπει αντίστοιχα να απευθυνθούμε στα αρμόδια όργανα και στου συναδέλφου που ασχολούνται με το Euromed. Μιλούν με βουλευτές από τη χώρα σα Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και τώρα των Α, μισό λεπτό, διότι έχουμε εδώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκπρόσωπό τη έχει να υποβάλει κάποιε παρατηρήσει. Οπότε θα πρέπει να δώσω το λόγο στον κύριο Αμύρ Μοταχάρη που είναι ο desk officer για Euromed και περιφερειακά θέματα ε, για την ρέλεξ της Κομισιόν. Συγγνώμη παρελίγο να σας ξεχάσω. Δεν το έκανε επίτηδες. Μουταχάρη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μας καλέσατε σε αυτή την δημόσια κρόαση. Άκουσα. Όλους τους έλαβαν το λόγο. Σαν όμορφη, γλυκιά μουσική είναι αυτά τα οποία άκουσα για την Αίγυπτο και για τον Μπαχρέιν. Είναι θέματα τα οποία τα ξέρουμε, μια που συνεργαζόμαστε με τους ε, εταίρους μας τις χώρες της Μεσογείου και υπάρχει ήδη ένα πλαίσιο εποπτείας, παρακολούθησης, συνεργασίας για πολιτικές μεταρρυθμίσεις, ανθρωπινά δικαιώματα σε σχέση και με τα προγράμματα δράσης. Αυτά όσον αφορά την επίσημη συνεργασία. Επί της ουσίας τώρα, επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει να πει ότι πρόσφατα και πιο συγκεκριμένα το 2009 έχουμε δει σε διάφορα ζητήματα πισωγύρισμα σε κάποιες χώρες. Χώρες που είχαν υψηλή προτεραιότητα τις μεταρρυθμίσεις, χώρες που ήταν πρωταθλητές, καλύτεροι μαθητές. χώρες που με την πρόοδό τους ασκούσαν πίεση στις άλλες χώρες. Έχουμε όμως ε, εκεί πισωγίσματα όσον αφορά τη ανθρώπινα δικαιώματα, τους ακτιβιστές, τους bloggers. Προσπαθούμε με ό,τι μέσα έχουμε όλα αυτά να τα αντιμετωπίσουμε. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία. Έχουμε επίσης ε, θεματικά εργαλεία και μέσα για συγκεκριμένες ατομικές περιπτώσεις και όσον αφορά τη συνεργασία την εκλογική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε πολιτική έχουμε αποστολές παρατήρησης αλλά βέβαια για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να μας καλέσει η σχετική χώρα. Επομένως, προς το να έχουμε μόνο δύο περιπτώσεις όπου ζητήθηκε τέτοια αποστολή. Πρώτα-πρώτα στα κατεχόμενα στην Παλαιστίνη και δεύτερη περίπτωση ήταν ο Λίβανος. Όσον αφορά την Αίγυπτο, προσφέραμε τέτοια αρρωγή, αλλά απερίφθη το αίτημά μας από την Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Τώρα, όσον αφορά τα δίκτυα και τις σχετικές δραστηριότητες, ανέφερε ο κύριος από την Αλγερία κάποιες αλλαγές που δεν ήρθαν από τα έξω, αλλά από τη βάση, από την κοινωνία. Έχουμε μια σειρά προγραμμάτων επίση για την ελευθερία των μέσων ενημέρωση, επικοινωνία, ε, εκπαίδευση δημοσιογράφων, τεχνική αρρωγή. Όμω, κάθε φορά είναι διαφορετικό ο συνομιλητή. Έχουμε κυβερνήσεις που στι περισσότερε περιπτώσεις είναι αυταρχικέ κυβερνήσεις. και σε σχέση με κάποια τεχνικά, τεχνοτικά θέματα, εμπορικά. Εκεί υπάρχει πρόοδος, αλλά όχι στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό τους το έχουμε πει, τους το έχουμε τονίσει. Το αναφέρουμε και στις εκθέσεις πρόοδο για το 2009 και για την Ισία και για Αίγυπτο, ακόμα και για το Μαρόκο. Τονίσαμε τους τομείς όπου υπήρχε σε Είναι μια δύσκολη, περίπλοκη γεωγραφική περιοχή. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά είναι γνωστοί οι κανόνες του παιχνιδιού. Τους ξέρετε, τους έχετε εγκρίνει εσείς. Είπαμε conditionality, αλλά θετική. Ερεσιμότητα θετική. Ερεσιμότητα είπαμε. Να επικριθεί, να συζητηθεί ο κανόνας του παιχνιδιού αυτός, αλλά είναι δεδομένος. Κάτι τελευταίο τώρα. Η διαφορά και η απόσταση μεταξύ του νόμου και του τι γίνεται στην πράξη. Πολλές φορές υπάρχει κλοκή νομοθεσία, υπάρχει ο κατάλληλος νόμος, αλλά δεν εφαρμόζεται στην πράξη. Υπάρχει μόνο αυτό το χάσμα μεταξύ πρακτικής και θεωρίας. Να ένα θετικό παράδειγμα. Έχει δημιουργηθεί η Ιορδανία. Να, πέρσι το αντιμετωπίσαμε αυτό. Όμως, ακόμα έχει δρόμο ο δημοσιολογητής αυτός, ούτως ώστε να μπορέσει να αποτελέσει ένα κοινωνικό γεγονός, πραγματικότητα. Να χωνέψει η κοινωνία τι είναι δημοσιολαβητής, τι αρμοδιότητες έχει, τι μέσα έχει στη διάθεσή του ως προς την κυβέρνηση και τη διοίκηση. <clears throat> Εν κατακλείδη, να σας πω ότι και εμείς δεν είμαστε τέλεια, και εμείς δεν τα έχουμε πάει παντού καλά, δεν έχουμε προσέξει τόσο πολύ τις κοινωνικές πολιτικές, τα κοινωνικά αιτήματα, εργασιακά, εργατικό δίκαιο, τις, ε, τα πρότυπα και τις ε, συμβάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Οπότε, έχουμε και τις πολυμερείς επαφές, ας πούμε θα κάνουμε την Υπουργική Σύνοδο τον Νοέμβριο, εδώ θα γίνει αυτό στις Βρυξέλλες. και έχουμε παραλήψει να προσέξουμε όσο πρέπει αυτούς τους κοινωνικούς εταίρους και τα αιτήματα της κοινωνίας. Σας ευχαριστώ κύριε Μουταχάρη, πάρα πολύ ενθαρρυντικά όλα αυτά όσον αφορά και την ε, ε, ένταξη της υπόθεσης ανθρώπινα δικαιώματα στη δική σας δουλειά, στα δικά σας θέματα. αυτό μας προσφέρει και στο μέλλον. πώ δηλαδή είναι δυνατόν η πολιτική των δικαιωμάτων να περάσει μέσα από τις επιμέρους πολιτικές τη ε, πολιτική γειτονία, τη ε, ευρωμεσογειακής ε, πολιτική και θα πρέπει η δική μας Επιτροπή να κάνει περισσότερες τις περισσότερα ταξίδια σε αυτές τις χώρες και ελπίζουμε να προχωρήσει αυτή η πρόταση. και ελέγχθη από τον υπόσχο της Συρίας ότι πήγαμε, σαντίσαμε τις αρχές της Συρίας, μιλήσαμε με αυτούς που είχαν φυλακίσει τον πατέρα του, ότι δήθεν είχε εξυβρίσει τις αρχές, των ε, πρόεδρο της χώρας και έτσι έχει καταρακώσει το ηθικό του λαού, λέγανε. Επομένω, πήγαμε στη φυλακή, τον είδαμε και ήταν πάρα πολύ σημαντικό το ότι προσπαθήσαμε να δούμε τι γίνεται, τι γίνεται αν υπάρχουν βασανιστήρια, τι γίνεται με το σοφρονιστικό σύστημα. Άρα, μπορούμε να πετύχουμε πράγματα αν είμαστε πιο δυναμικοί, να απευθυνθούμε και στο Συμβούλιο του ΟΗΕ, το αρμόδιο, και τις επόμενες ε, συναντήσεις μας θα έχουμε την ε, παρουσίαση της έκθεσης του ΙΕ για τις μυστικές φυλακές, τα μυστικά στρατόπεδα περιορισμού που υπάρχουν στον κόσμο. Τώρα, να δούμε ποιες να δούμε το λόγο. Πρώτος ο κύριος Ομπιόλς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα ακούσαμε για πολύ συγκεκριμένα θέματα. Έχω κάτι να πω σαν παρατήρηση και κάποιες ερωτήσεις. Έχω να παρατηρήσω το ότι η δυτική οπτική και όχι μόνο ευρωπαϊκή, η δυτική μια που λέμε και για το Freedom House όσον αφορά τον αραβικό κόσμο πολλές φορές ε, ε, κάνει το λάθος το να ε, τους βάζει όλους στο ίδιο καζάνι, στο ίδιο καλάθι, στον αραβικό κόσμο ας πούμε. Γιατί υπάρχουν διαφορές από χώρα σε χώρα και λόγω καθεστώτων και λόγω θεσμών ε, και λόγω κοινωνιών τα πράγματα διαφέρουν μια χώρα στην άλλη στον αραβικό κόσμο και γι' αυτό σας λέω είχαμε πάρα πολύ διαφορετικές αποχρώσεις όσα ακούσαμε πούμε, από τον κύριο Μπουμαλά και από τον κύριο Σαντάτ φάνηκαν οι, οι διαφορές αν κατάλαβα καλά ο κύριος Σαντάτ βλέπει τον εκδημοκρατισμό και την κατάσταση των δικαιωμάτων σε πρώτη χώρα του σαν κάτι πάρα πολύ σημαντικό ως αναγνώριση μιας πραγματικότητας πολιτιστικής, θρησκευτική, οργανωτικής μέσα και από την, την, παράδοση που, έχουν οι, που έχει η μουσουλμανική αδελφότητα. Θεωρεί ότι είναι ακρογωνίως λίθος αυτός για τον δημοκρατικό μετασχηματισμό της χώρας. Το ενώ ο κύριος Μπουμαλά μας τα έλεγε κατά στον τρόπο διαφορετικά ότι δηλαδή Μετά τον εμφύλιο πόλεμο, μετά αυτή την τραγωδία, υπάρχει μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Από από το φόβο του, το, το να γίνει πάλι κάτι τέτοιο. Διάλογος, συνεννόηση. Μεταξύ αυταρχικής εξουσίας και του ζωσπαστικού Ισλαμικού κινήματος. Έχουμε από μέσα εδώ πέρα δύο διαφορετικές οπτικές που αυτό μας δείχνει το ότι δεν θα πρέπει να γενικεύουμε. να μην γενικεύουμε ούτε και για το θέμα της από, της τα μέσα αλλαγής μεταρρύθμισης. Θα πρέπει να λαμβάνει την υπόψη ρυθμίες κάθε χώρας. Η ερώτηση τώρα προς τους συνομιλητές μας έχει να κάνει με κάτι το οποίο είπε τα κ με τον οποίο συμφωνώ. Και για την αιρεσιμότητα ιδίω. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και θα πρέπει να δίνουμε κίνητρα. Μας μίλησε τα χάρη για πίσω γύρισμα σε αυτές τις χώρες. Πολύ σημαντικό αυτό. σύμφωνοι. Όπως και να η κατάσταση μια χώρα, είτε είναι κακή, είτε μέτρια, είτε καλή, το θέμα είναι τι, τι, τι τάση υπάρχει. Τάση για βελτίωση, τάση για επιδείνωση. Βέβαια, ακριβώς, άμα κανείς θεωρήσει ότι είναι σε καλή κατάσταση και τα πράγματα επιδεινώνονται, αυτό είναι κακό. Ή ε, αντίστροφα, εάν η κατάσταση είναι κακή και τα πράγματα βελτιώνονται, τότε τα πράγματα είναι αισιόδοξα. Στη ΔΕ Αίγυπτο Έχουμε εξελίξεις. Γίνονται πράγματα. Όπως ε, υπενθυμίστηκε, το 2011 θα έχουμε εκλογές. Και ε, αυτή η προσωπικότητα πολύ προβλημένη στη Δύση πρόκειται να κατέβει σε εκλογές που έχει το ειδικό βάρος για να μπορέσει να συσπυρώσει μεγάλα κομμάτια, μεγάλους τομείς της ε, κοινωνίας και των, της μεσαίας τάξης. Μα ακριβώ αυτό που είπατε και εσεί κύριε Σαντάτ. Όσον αφορά την μουσουλμανική αδελφότητα. Εσείς τι προγνωστικά κάνετε. Πάμε προς χειρότερα ή υπάρχει ελπίδα στο μέλλον. Αλγερία είχαμε έναν διπλωμάτη που όταν είχαμε αυτή την τρομερή σύγκρουση είχαμε μια κατάσταση πάρα πολύ στατική και προχωρήσαμε προς μια φάση όπου βρισκόμαστε σε προσδοκή εξελίξεων αλλά και εκεί πέρα δεν ξέρω κύριε Μπουμαλά τι λέτε εσείς τι προγνωστικά κάνατε πώς τα βλέπετε όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα Ευχαριστώ κύριο Μπιόλς Τώρα θα δώσουμε το λόγο στους τρεις ομιλητές μας σύντομα να δώσουν απαντήσεις. Όλοι είστε προσκεκλημένοι σε μία μικρή reception, την οποία οργανώνουμε μαζί με το Freedom House, για να υπογραμμίζουμε την σημαντική προσπάθεια την οποία κάνουν οι νέοι ακτιβιστές στις χώρες αυτές. Κύριε Σαντάτ, κάποιες ερωτήσεις σαν για σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το ότι στην Αίγυπτο έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος. Αν και η πρόοδος αυτή δεν είναι επαρκής. Χρειάστηκε πολύς χρόνος για να υπάρξει και θεωρούμε ότι από τις ε, τελευταίες εκλογές του 2005 όλοι είχαμε πολλές ελπίδες να υπάρξει περισσότερη πρόοδος, περισσότερες δυνατότητες για τον πολιτικό κόσμο, αλλά δυστυχώς όμως πήγαμε και εκεί προς τα πίσω. Όταν η κυβέρνηση είδε την επιτυχία των μουσουλμάνων αδελφών, 88 έδρες, ανησύχησε. Ξέρετε ότι οι εκλογές μας γίνονται σε τρεις φάσεις και γι' αυτό στη δεύτερη και στην τρίτη φάση στην ουσία έκαναν τη ζωή δύσκολη για όλους τους υποψηφίους στη δεύτερη και στην τρίτη εκλογική αναμέτρηση. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε είναι να πείσουμε ότι η Αίγυπτος αξίζει να βρεθεί σε μια καλύτερη